Hi. Good morning. Καλημέρα σας. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Καλημέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Καθίστε παρακαλώ. Πρώτο σημείο έχουμε την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. έχουμε κάποιες ε, αλλαγές πιο συγκεκριμένα στο σημείο 15 την αντιπροσωπεία της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στην Αθήνα και ζητήθηκε να αναβληθεί για τη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου. Αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι την η μερίσια διάταξη με την αλλαγή την οποία σας ανέφερα. Σημείο 2. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Θα σας διαβάσω τις ανακοινώσεις στα αγγλικά, γιατί οι σημειώσεις που έχω εδώ είναι στα αγγλικά. Έχουμε ένα διορθωτικό έγγραφο το οποίο θα ε, προσθεθεί στο κείμενο για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Εγκρίθηκε ο κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου και δεν ε, συμπεριέλαβε και τα αποτελέσματα της επαλήθευσης που γίνεται από τους γλωσσομαθείς νομικούς. Έχει λοιπόν να διανεμηθεί ένα διορθωτικό έγγραφο ε, γιατί θα υποβληθεί στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου βάσει του άρθρου 216 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εάν δεν υπάρχει κάποια ένσταση μέχρι το πέρας της συνεδρίασης, ε, θα θεωρηθεί ότι εγκρίνεται το διορθωτικό αυτό κείμενο, το corrigendum, και θα περάσει επευθεία στην Ολομέλεια. Σημείο Β. Δεν υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν χρησιμοποιήθηκε η διερμηνία ή καθυστερημένες ακυρώσεις από την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης. Σημείο Γ, web streaming και ε, το αρχείο των ηλεκτρονικών συνεδράσεων. Όλα αυτά είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-meeting και οι συνεδρίες φυσικά μεταδίδεται μέσω web streaming στο διαδίκτυο. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 3 και θα περάσω και πάλι στα πορτογαλικά. Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2012. Γνωμοδότηση. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης είναι ο κύριος Άνταμ Κόσα. Και του δίνω απευθείας το λόγο. προκειμένου να μας παρουσιάσει τις συμβιβαστικές τροπολογίες ε, τις οποίες συζητούμε επί του θέματος. Köszönöm szépen a szót, Kedves kollégák, úgy gondolom, hogy... Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι ήταν υποδειγματική η συνεργασία μας το θέμα αυτό. Βεβαίως και υπήρξαν κάποιες ε, αποκλήσεις, στις απόψεις μας, αλλά καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια εξαιρετική συμφωνία ε, με τις συμβιβαστικές αυτές λύσεις. Έχουν κατατεθεί δύο συμβιβαστικές τροπολογίες. διότι δεν καταφέραμε να τα συμπεριλάβουμε όλα σε μία συμβιβαστική τροπολογία. Επομένω, έχουμε δύο συμβιβαστικέ τροπολογίε, την Α και τη Β. Όσον αφορά τη συμβιβαστική τροπολογία Α, Συγγνώμη, μισό λεπτό να βρω και πού είναι και το σημείωμα. Η κυρία Δίπελ και η κυρία Λάμπερτ υπέβαλαν τροπολογίες και καταλήξαμε σε μια συμβαστική λύση την οποία υποστηρίζουν και οι δύο συνάδελφοι. Έτσι καταφέραμε να έχουμε ένα κείμενο το οποίο ε, μπορεί να συμπεριληφθεί στο υπόλοιπο κείμενο. Όσον αφορά τη συμβαστική τροπολογία Β, ακολουθήσαμε την ίδια διαδικασία. Υπάρχουν εδώ όμως δύο δυσκολίες και θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας σε αυτές τις δυσκολίες. Η πολιτική μου ομάδα δεν υποστηρίζει κάποια στοιχεία των τροπολογιών διότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες με τις οποίες δεν μπορώ να συμφωνήσω. Τι ακριβώς εννοώ. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε από την πρόεδρο της Επιτροπής μας και ε, βάσει αυτού να σας πω ότι υπάρχει ένα αρχικό κείμενο το οποίο είχα αποβάλει πριν από δύο μήνες και βάσει αυτού του αρχικού κειμένου την προηγούμενη εβδομάδα με ενημέρωσε η πρόεδρος ότι διαγράφεται μία παράγραφος. διότι η παράγραφος αυτή δεν είναι της αρμοδιότητας της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Δεν αμφισβητώ βέβαια σε καμία περίπτωση την, ε, τις γνώσεις Προέδρου και το γεγονός ότι είναι αρμόδια από αυτού του θέματος, απλώς δεν καταλαβαίνω γιατί σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας ε, γίνεται αυτή η αλλαγή. Καταφέραμε βέβαια να καταλήξουμε σε ένα καλό συμβιβασμό θεωρώ και μέχρι την ψηφοφορία του κειμένου είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε επί ενός κειμένου το οποίο θα μας επιτρέψει να δώσουμε ένα καλό προσανατολισμό στην αρμόδια επί επιτροπή, στην Επιτροπή ε, Πολιτικών Υποθέσεων, Πολιτικών Ελευθεριών. Να σας πω ότι το κείμενο αυτό άπτεται της κατάστασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων το 2012. Μπορεί βέβαια να υπάρχει διάσταση απόψεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα τη σήμερα ημέρα και γι' αυτό ακριβώ είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, τα δικαιώματα που αφορούν τον κοινωνικό τομέα να συζητηθούν και αυτά και να ε, συμπεριληφθούν και αυτά στα βασικά κείμενα και να λαμβάνουμε υπόψη και τις συνθήκες και τα βασικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω ότι όλα αυτά τα έχουμε λάβει δεόντως υπόψη και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ah, Ευχαριστώ κύριε Κώσα. Η κυρία Ζήπλα έχει ζητήσει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μπορώ να είμαι και σύντομη. Ήδη στην προηγούμενη συνεδρίαση αναφέραμε ότι δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην έκθεση αυτή. Μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον συμβιβασμό αυτόν. Έχουμε πετύχει καλό αποτέλεσμα και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιδιαίτερα με τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων. Νομίζω ότι είναι καλή η έκθεση στην οποία έχουμε καταλήξει. Υπάρχουν διστάμενες απόψεις για κάποια σημεία, αλλά Ιδιαίτερα με τις συμβαστικές τροπολογίες έχουμε καταλήξει σε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να ε, ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορώ να είμαι παρούσα στην ε, ψηφοφορία διότι έχω έκθεση σε άλλη επιτροπή αλλά είμαι βέβαιη ότι θα πετύχουμε καλή πλειοψηφία για την έκθεση αυτή, υπέρ της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κώσα για την δουλειά που έκανε. Ήταν στη διάθεσή μας για να συζητήσουμε ε, διάφορα θέματα ε, πολύ συχνά και είμαι ευγνώμων γι' αυτό όσον αφορά την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής μας πάνω στην έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το αρχικό σχέδιο ε, περιείχε πολύ λίγα στοιχεία δικά μας. Η έκθεση ΛΥΜΠΕ είχε καλυφθεί στο σύνολό της, αλλά η δική μου συνεισφορά καθώς και άλλων ε, δεν είναι στην έκθεση. Η Άλτη στηρίζει το μεγαλύτερο μέρος των τροπολογιών και τις ε, συμβαστικές τροπολογίες, αλλά υπάρχουν ακόμα κάποια προβληματικά σημεία. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την τροπολογία 17. Δεν είναι η Τρόικα υπεύθυνη για τις ε, δυσκολίες που αντιμετωπίζουν διάφορες χώρες και όσον αφορά την 11 και την 12 θα απόσχουμε από την ψηφοφορία διότι δεν πιστεύουμε ότι ταιριάζουν με το υπόλοιπο του κειμένου. Στην ε, περίπτωση της τροπολογίας 11 και τις 12 ε, ε, είναι αρκετά ασαφής, δεν είναι αρκετά ακριβής. Όσον αφορά την τροπολογία 20. Θα θέλαμε εξοχωριστή ψηφοφορία στο σημείο αυτό δεν υπάρχουν όμως σημαντικά προβλήματα με το έγγραφο αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κόσα για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει και η Άλντε θα υπερψηφίσει τη γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Οβίρ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στην Κομισιόν. Έχετε παρατηρήσεις για την έκθεση αυτή? Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Κύριε Σιγητά, θέλετε κάτι να συμπληρώσετε? Ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις παρατηρήσεις και εγώ θεωρώ ότι ο στόχος ήταν κοινός και έχουμε όμως μια διαφορετική προσέγγιση ως προς το στόχο. Εγώ εργάστηκα υπό το πνεύμα της Χάρτας των Θεμολογικών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβα επίσης υπόψη και τις ε, διαδικασίες της Επιτροπής ΛΥΠΕ. Όσον αφορά την τροπολογία 17, η πολιτική μου ομάδα δεν την υποστηρίζει και δεν θα υποστηρίξουμε επίσης και την τροπολογία 22. Για τις υπόλοιπες τροπολογίες και τις προφορικές τροπολογίες, αυτές τις υποστηρίζουμε όλες και νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα καλό κείμενο. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά τη διαδικασία που ακολούθησε η Πρόεδρος, ε, της Επιτροπής μας, αποφάσισα να αποφασίσω ευθύ εξ αρχής τι πρέπει να γίνει, διότι αν έχουμε διαφορετική άποψη για τις διάφορες τροπολογίες θα διευκολυνθούν καλύτερα οι εργασίες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κώσα. Η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα εδώ στην Επιτροπή Απασχόλησης, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί 16 ή 17 Δεκεμβρίου. Και υπολογίζουμε τον Ιανουάριο να ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Okay. Tenho a informação Με ενημερώνουν ότι η εισηγήτρια για το επόμενο θέμα, το σημείο 4, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για τη διοργάνωση δειγματοληπτικής έρευνας ε, σχετικά με το εργατικό δυναμικό στην κοινότητα, δεν είναι παρούσα. Α, και όμως μου λένε. Μόλις, μόλις έφτασε. No, she's not here. She's not here. Ε, Peço desculpa. Parece que de facto a relatora não está presente na sala. Zito, Ζητώ συγγνώμη, όχι, δεν είναι παρούσα. Λάθος με ενημέρωσαν. Τρία λεπτά διάλειμμα και θα περιμένουμε να καταφτάσει η συγκήτρια. Chers collègues, il est 9h33. Αγαπητοί συνάδελφοι, 9.33, 3 λεπτά καθυστέρηση, συγγνώμη. Παρακαλώ καθίστε. Να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες με το 5, την ψηφοφορία για την έκθεση πρωτοβουλίας την κοινωνική προστασία για όλους και για τους αυτοαπασχολούμενους. Πρόκειται για έκθεση όπου η κυρία Βίντσελη Τσουτέ ήταν η, η και έχουμε και μια γνωμοδότηση της Επιτροπής Γυναικών. Για το τμήμα 1. Έχετε όλοι και τον υπότιτλο ένα μάλλον καλύτερα. Αλλά ο κύριος Μπένιον, Άνιον. Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν κάποιες συμβαστικές τις οποίες δεν υποστηρίζουμε όπου αναφέρεται το όνομά μας. Για να το έχετε υπόψη σας όπως θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. γιατί οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν μέχρι αργά χθε το βράδυ. Πολλοί συμβιβασμοί που αναφέρονται ότι υποστηρίζονται από εμά δεν υποστηρίζονται από εμά, αλλά δεν είναι πρόβλημα. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όλοι περί τίνο πρόκειται. Ποιε είναι παρακαλώ αυτέ οι τροπολογίε ή να σα ρωτάω κάθε φορά. Όχι, όχι. DHJ S V και ΑΑ. DHJ, XV και ΑΑ. Ωραία λέει πρόεδρος. Εντάξει, αν το πω είναι λάθος. Αν πω ότι υποστηρίζετε αυτέ τι τροπολογίε είναι λάθος όπω τα διαβάζω. Λοιπόν, υπότιτλος 1, ε, τροπολογία 35, Μπέκερ, υπέρ. Κατά αποχές, λοιπόν, πρώτη ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 13 υπέρ, 14 κατά, 3 αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 1. Συμβαστική I. Από 4 ομάδες. Και η φιλελεύθερη. είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 1. Συμβαστική J. Από 3 ομάδες. Υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Ε, η τροπολογία 6 της Επιτροπής Γυναικών, η συγκιτρια υπέρ υπέρ. Εγώ βλέπω υπέρ ότι είναι η συγκίτρια Α, άλλαξε γνώμη η συγκίτρια Λοιπόν, άλλαξε γνώμη η συγκίτρια αλλά δεν είναι εδώ στο κατάλογο ψηφοφοριών. Δεν είναι σοβαρά αυτά. Εν πάση κατά η συγκίτρια υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 της Επιτροπής Γυναικών, η συγκιτρια υπέρ, άλλη υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 42. Καταπίπτει. Παράγραφος 3. Συμβαστική κάπα από 4 ομάδες υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 3. Συμβαστική αβ. 4 ομάδων υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Συμβιβαστική L. 4 ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 4. Τροπολογία 1 της Επιτροπής Γενικών Ισχύτρια υπέρ. Α, όχι, είναι κατά. Άλλαξε άποψη. Οι γυναίκες αλλάζουν ε, γνώμη. Κατά αποχές απορρίπτεται. Όχι, οι γυναίκες δεν αλλάζουν άποψη. Καλά. Τροπολογία 3 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 5 συμβαστική μη από τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 5, συμβαστική νη τεσσάρων ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12, η συγκίτρια είναι υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 της ίδιας επιτροπής. Υπέρ η συγκίτρια υπέρ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε. Νομίζω ότι καταπίπτει. Όχι, ε, μάλλον ότι απορρίπτεται νομίζω. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. 15-16 απορρίπτεται. Μηδέν αποχές. Τροπολογία 14. Γυναικών εισηγήτρια υπέρ, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Γυναικών εισηγήτρια υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Γυναικών υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 γυναικών, η είναι κατά υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 6, συμβαστική όμικρον 4 ομάδων υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 7, συμβαστική π 4 ομάδων υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 7, τροπολογία 8 της Επιτροπής Γενικών Υπέρ αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q, 4 ομάδων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8 συμβαστική ρο ε, υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική S 4 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παραφωνία, 9 τροπολογία 84 της εισηγήτριας με προφορική τροπολογία της ομάδας Άλντε. Υπάρχει καμία αντίρρηση στην προφορική τροπολογία όχι. Ωραία ψηφίζουμε την τροπολογία 84 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Παράγραφο 13, τροπολογίε απάλληψη, οπότε θα ψηφίσουμε τη συμβαστική ΤΑΦ τεσσάρων ομάδων. Είναι οι τροπολογίε 85 Εσαγιά, 86 Μπέκερ, 87 ΜΑΝΑ. Ποιοι είναι υπέρ αυτών των τριών τροπολογιών. Κατά αποχέ απορρίπτονται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική ΤΑΦ τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Μετά τη 10, συμβαστική ΙΟΥ 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 11.2. απαλληπτικές 93. Εσάγια 94. Σόγκορ. Υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Ελέγχουμε τις απαλληπτικές τροπολογίες. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Με 15-16 απορρίπτονται. Μετά την παραφορά 11. Τροπολογία 95. Καταπίπτει. Περνάμε στην τροπολογία 96. από δύο συναδέλφους των Πρασίνων, όπου έχει ζητηθεί κατά τμήματα ψηφοφορία από την Άλδε, Πρώτο τμήμα, χωρίς τις λέξεις ε, με τη μορφή ε, ενός κατώτατου ορίου κοινωνικής προστασίας στην Ένωση. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές, να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 96. Άρχεται, ψηφίσατε πέρας. Με 19-12 εγκρίνεται. Ψηφίζουμε λοιπόν το δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε και εδώ έλεγχος του δεύτερου τμήματος. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ισοψηφία 16 απορρίπτεται. Παράγραφος 13, απαλληπτικές 97 έως 99, τον Εσαγιάμαν Σόγκορ, οπότε θα ψηφίσουμε τη ΒΕΑ αν εγκριθούν, που, από τριών ομάδων ποιοι είναι υπέρ της απάλληψης, της 12. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Β, τριών ομάδων υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Μετά τη 13, τροπολογία 102, Μπεναγάμπα Του και Κορνέλισεν, ποιοι είναι υπέρ κατά Αποχές να ελέγξουμε. Την 102 άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Ισοψηφία 16 απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 103 εσαγιά. Συγκήτρια κατά. Υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Της 103. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 16 υπέρ 11 κατά 5 αποχές εγκρίνεται χάρη τις αποχές μετά την παράγραφο 13 τροπολογία 104 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε να ελέγξουμε την 104 Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας, 19 υπέρ, 13 ε, κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Ε, τροπολογία 105 του ιδίου συντάκτη υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την 105 άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας, ισοψηφία 16 υπέρ 16 κατά, απορρίπτεται. Παράγραφος 13, συμβαστική τροπολογία έρφαση υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 14, συμβαστική W, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15, 110 σαρίες αγιά, από ε, διαγραφή, ε, συμβαστική X, γιατί 10, 110 ε, λοιπόν απορρίπτεται, X από τρεις ομάδες υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 16. 115 πάλι διαγραφής από την Εσαγιά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ή ε, από τρεις ομάδες υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Μετά παράγραφος 10 Επιτροπή Γενικών Υ. εισηγήτρια είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17Z από τρεις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 παράγραφος. Οι 128 και 129 καταπίπτουν. Παράγραφος 18 συμβαστική ΑΑ από τρεις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18-133 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να κάνουμε μια παλήθευση για την 133, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 14 κατά, καμία, 3 αποχές. Εγκρίνεται. 18, 136. Μπεναρά του Κορνέλισεν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Καταπίπτουν όλες οι τροπολογίες και πάμε στην 20. Καταπίπτουν επίσης όλες. Αιτιολογική σκέψη α, συμβιβαστική α, τέσσερις ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 Μπένιον, κατά η εισηγητρία υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Για την τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 12 κατά, μία αποχή, εγκρίνεται. Με μεγάλη διαφορά. Ε, Τιολογική σκέψη Β, συμβαστική Β, από τρεις ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική σε από τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε αιτιολογική σκέψη ε τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά, παράγραφος α της Επιτροπής Γυναικών, υπέρ εισηγήτρια, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Β της ίδιας επιτροπής υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Σ της ίδιας επιτροπής υπέρ, επαλήθευση για τη Β. Παράγραφος Β της Επιτροπής Γυναικών. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 17 κατά. Ισοψηφία. Καμία αποχή. Απορρίπτεται. Παράγραφος Σ της ίδιας Επιτροπής υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση για τη ΣΥ, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρασε ψηφοφορίας, 21 ψήφοι υπέρ, 13 κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν σαφέστατα. Παράγραφος D της Επιτροπής Γυναικών υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος ε της Επιτροπής Γυναικών υπέρ, κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται να το επαληθεύσουμε όμως άρχεται η ψηφοφορία θα δούμε, θα δούμε, περιμένετε Πέραση της ψηφοφορίας 17-14 3 αποχές εγκρίνεται αιτιολογική F συμβαστική F από Τέσσερις ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 25 του κυρίου Πουπάκη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 26 του ίδιου συντάκτη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική G. Τροπολογία 27 που είναι ε, διαγραφή από την Σαρία Σεγιά υπέρ της διαγραφής κατά, αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική τροπολογία G από τέσσερις ομάδες, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, κλείνει το μικρό. Τροπολογία 30, για Γεσλοπιέσκα, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος F της Επιτροπής Γυναικών, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική H, από τέσσερις ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ολοκληρώσαμε με τις τροπολογίες και να ψηφίσουμε λοιπόν το σύνολο του κειμένου με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Tout monde a pu voter, le vote est clos. Ψήφισαν όλοι, πέρα ψηφοφορία, 29 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, μία αποχή, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια.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 ε, αρμόδια η Επιτροπή μας και ήταν και η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων αρμόδια για το θέμα το. Η τροπολογία 90 της κυρίας Τάουνμπουργκ, αν δεν κάνω λάθος, έχει αποσυρθεί. Στον κατάλογο ψηφοφοριών η Ευρώπη των Συντηρητικών και Δημοκρατών δεν υποστηρίζει τις ε, συμβαστικές τροπολογίες D, R και V. Και για την τροπολογία 11 της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων έχουμε μία προφορική τροπολογία την οποία έχει παρουσιάσει η Ομάδα των Φιλελευθέρων. Προτείνω λοιπόν να συζητήσουμε την προφορική τροπολογία όταν θα φτάσουμε στην ε, ψηφοφορία ε, σύμφωνα με τη σειρά. Κύριε Σιγητά, σχόλιο εκτός μικροφώνου, να πάρετε το λόγο όταν θα φτάσουμε στην τροπολογία αυτή. Ε, Παράγραφος 1, τροπολογία 40, Σάρια Σάγια. Κατά ο συγητή υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 4 τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πριν συνεχίσουμε με την ψηφοφορία, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι βάσει του άρθρου 50 δεν θα ψηφιστεί παρά, ε, ψηφιστούν παράγραφοι 3, 9, 10, 12 και 13 της Επιτροπής ΕΚΟΝ, διότι πρόκειται για θέματα στα οποία έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα και επομένως ε, θεωρούνται ήδη εγκεκριμένα. Παράγραφος 2, συνεχίζουμε, 41, εσάρια σε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε την παράγραφο 6 της ΕΚΟΝ, υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται νομίζω, αλλά να κάνουμε μια επαλήθευση. Για την 6 της έκον. Παράδοξα πράγματα. 12 υπέρ, 21 κατά. Απορρίπτεται. Παράγραφος 3. 42 σάριες Άγιο υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση για τη 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρασε της ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται. Παράγραφος D, συμβιβαστική τροπολογία από 5 ομάδες το ECR απέσυρε την υποστήριξή του υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μεγάλη αγωνία. Μετά την παράγραφο 4, παράγραφος 5 της ΕΚΟΝ, υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Για την 5, νομίζω ότι απορρίπτεται. Ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 17 κατά, απορρίπτεται. Μετά, τροπολογία 53 της Αρίας Άγια, η συγκεκριμένη κατά υπέρ. Τι πρόβλημα υπάρχει. Δεν έχω μια σελίδα νομίζω, είμαι βέβαιη ότι μου λείπει μια σελίδα από τις ψηφοφορίες. Ε, δεν έχω, λείπει μια ολόκληρη σελίδα. Εσείς είστε σε καλύτερη κατάσταση από μένα. Παπαπα. 8 έκον υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την 8. Nous 8 de la Commission économique monétaire. Le vote est ouvert. 8 της ΕΚΟΝ. Άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι. 20 υπέρ, 15 κατά, εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Τροπολογία 45, Σαρισάγια, υπέρ. Κατά, αποχές Η 46 Ρέγνερ είναι συμβατή σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα χωρίς τον όρο National υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και την προσθήκη του όρου National τώρα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 5 2 της ΕΚΟΝ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα χωρίς το issue as a type of deferred compensation για το υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Προστίκη αυτής τη φράση υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 15 της ΕΚΟΝ υπέρ, κατά αποχές επαλήθευση. Για τη 15 της ΕΚΟΝ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 15 κατά. Εγκρίνεται. Με τρεις αποχές. Παράγραφος 6, συμβιβαστική τροπολογία J. Από 5 ομάδες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 7, συμβιβαστική τροπολογία K. Από 5 ομάδες υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7, το 93 Σάρι Σάγια, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 8, δύο τροπολογίες για διαγραφή, 54 Εσάγια και 55 Γιούτα Στάιρουκ, είναι κατά ο εισηγητής υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Παράγραφος 8, συμβαστική τροπολογία L από τέσσερις ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 8, συμβαστική τροπολογία M από 5 ομάδες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 8, 11 της Επιτροπής ΕΚΟΝ και ο εισηγητής θα ήθελε εδώ να παρουσιάσει μια προφορική τροπολογία και θα ψηφιστεί και κατά τμήματα η τροπολογία. Αν κατάλαβα καλά, η προφορική σας τροπολογία είναι για το πρώτο τμήμα. Έχετε το λόγο. Ναι. Το δεύτερο τμήμα, από ό,τι κατάλαβα, δεν θα ψηφιστεί. Το πρώτο τμήμα, η προφορική τροπολογία λέει believes that an impact assessment, προσθέτουμε δηλαδή και το an impact assessment στη φράση, για να εξετάσουμε με ποιος τρόπο θα έχουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού και θα αποφύγουμε την παρακόλληση της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων. Έτσι, η τροπολογία αυτή ευθυγραμμίζεται με τις συμβασμούς που κάναμε, διότι συνεχώς αναφερόμαστε σε αυτή την αξιολόγηση των επιπτώσεων. Ενίσταται κάποιο στην τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα τη τροπολογία ΕΚΟΝ 11 Ω τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Με επικοδομητικές εποχές, λέει ο Πρόεδρος. Παράγραφος 14 της ΕΚΟΝ υπέρ. Κατά αποχές, επαλήθευση για τη 14. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 18 pour. Λοιπόν, πέρα προφορίε 18 υπέρ 16 κατά, 0 απόχέ. εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Δύο τροπολογίες απάλληψης. 62 Εσαγιά, 63 Ρέγνερ. Η συγκίτρια κατά υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Παράγραφος 10. Δύο τροπολογίες απάλληψης των ιδίων. Η συγκίτρια είναι κατά. Γιατί αν ψηφιζόταν δεν θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε τη συμβαστική εν τεσσάρων ομάδων. Ποιοι είναι υπέρ της απάλληψης. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική εν τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά ας ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. 22 υπέρ 13 κατά 0 αποχές απορρίπτονται μετά την παράγραφο 10 α όχι όχι εγκρίνεται νομίζω, εγκρίνεται ωραία μετά την παράγραφο 10 τροπολογία 7 της έκον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Στην παράγραφο 11, το εισαγωγικό τμήμα, συμβαστική όμικρον, πέντε ομάδων υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Στην παράγραφο 11, στο σημείο α, συμβαστική π, π, πέντε ομάδων υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Στο σημείο B, συμβαστική Q, πέντε ομάδων υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Για το σημείο C, η τροπολογία 15 ε, σαρίσα για υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, απορρίπτεται. Στο σημείο D, τροπολογία 76 της ίδιας, η συγκίτρια είναι επίσης κατά υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται. 77 Ρέγνερ για το ίδιο σημείο υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 11, στο σημείο E, συμβαστική άρα όπου ε, δεν ε, το, τη στηρίζει πλέον η ECR, οι άλλοι τέσσερι ναι υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Στο σημείο F, συμβαστική S, από πέντε ομάδες υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Στο σημείο G, συμβαστική TAF, πέντε ομάδων υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. Μετά το σημείο G, τροπολογία 86, Ρέγνερ, η συγκίτρια κατά υπέρ κατά αποχές Ωραία, δεν βλέπω να ψηφίζετε. άρα πρέπει να ελέγξω ηλεκτρονικά. Άρχεται για την 86. Ψηφίσατε όλοι πέρα. 17 επέρ 16 κατά. Δύο αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 87. Κάστλερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88. Ρέγνερ υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται ψηφίσατε όλοι Πέρας. 20 υπέρ 14 κατά μία αποχή εγκρίνεται 89 της ιδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παύλα 1. Συμβαστική τροπολογία. Α. Με συγχωρείτε, αλλά ε, δεν μπορώ να παρακολουθήσω το κατάλογο ψηφοφοριών, δεν το κάνω συνήθω. Παράγραφο 12. Έχει αποσυρθεί 90, οπότε ψηφίζουμε τη συμβαστική U. 5 ομάδων υπέρ κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται μετά την παραγραφό 12. Τροπολογία 1 έκον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 της ιδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 έκον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 13. Συμβαστική Β. Τεσσάρων ομάδων. Χωρίς τους συντηρητικούς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική αναφορά η τροπολογία 2 του εισηγητή υπέρ κατά εγκρίνεται. Η ίδια τροπολογία 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. Μετά την αιτιολογική αναφορά 14 3 Ρέγνερ υπέρ κατά εγκρίνεται. Στην αιτιολογική σκέψη α το εισαγωγικό τμήμα τροπολογία 4 Ρέγνερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ετελογική σκέψη α. Συμβαστική α. Τριών ομάδων. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ετελογική α. Εδάφιο 2B από πέντε ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε, μετά την ιδεολογική σκέψη α, έχουμε την τροπολογία 11, Ρέγνερ έπειτα της οποίας ωστόσο η ομάδα Άλντε έχει μία προφορική τροπολογία. Μα πώς είναι να τον έχουμε δύο τροπολογίες 11. Α, ήταν εικόνα 11 η προηγούμενη. Καλά. Ο συγητής θέλει να κάνει προφορικές τροπολογίες στο 11. Παρακαλώ κύριε συγητή, εξηγήστε μας αυτή την προφορική τροπολογία, γιατί την είχατε κάνει, είχατε κάνει προφορική τροπολογία στο άλλο 11. Μα δεν χρειάζεται να το εξηγήσω, το λέει το κείμενο. Όλοι γνωρίζετε λοιπόν αυτή την προφορική τροπολογία, δεν υπάρχει αντίρρηση, εγκρίνεται. Όχι, όχι θα, θα την ψηφίσουμε παρόλα αυτά. Τροποποιημένη 11 υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Αιτιολογική σκέψη Β, τροπολογία 12, εισαγιά, υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται μετά την αιτιολογική β. Τροπολογία 13 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ετυλογική σε σκέψη. Συμβαστική Σ, πέντε ομάδων και η συντηρητική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ετυλογική σκέψη D. Συμβαστική ε. πέντε ομάδων υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οπότε, μετά την ολογική D έχουμε τροπολογία 22 μπένιον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ε, συμβαστική F, 5 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη F, συμβαστική G, 5 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη G, συμβαστική H, 5 ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά την ειδική σκέψη H, τροπολογία 32, McIntyre, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ειδική σκέψη I, συμβαστική I, πέντε ομάδων, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οπότε, μετά την ειδική σκέψη I, τροπολογία 35, εισηγείται υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εταιρική σκέψη J, τροπολογία 36, Regner, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ετυλογική σκέψη Κ, τροπολογία 37, εσαγιά, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οπότε περνάμε στην τροπολογία 38, Μάκιντάιρ, υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να ελέγξουμε. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 17 υπέρ, 15 κατά, 3 αποχές. Εγκρίνεται. Μετά την ελογική κάπα, τροπολογία 39, Jean Lambert, με προφορική τροπολόγηση. Τη ομάδα ALDE, δεν υπάρχει αντίρρηση να υπάρξει προφορική τροπολόγηση, είναι τεχνικής φύσης, ψηφίζουμε τροπολογία 39, υπερκαταποχές, εγκρίνεται. Ωραία. Ψηφίσαμε τις ε, τροπολογίες. Ψηφίζουμε το, τροπο, το, το τροπεπιθέν κείμενο ηλεκτρονικά έρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 32 υπέρ, 3 κατά, 0 αποχές. Συγχαίρουμε τον εισηγητή. Περνάμε στο σημείο 7, κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για γνωμοδότηση. Αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή είναι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και ο συντάκτης είναι ο κύριος Κόζα. Πριν από την παράγραφο 1, τροπολογία 1, συγγνώμη, πρώτη παράγραφος 1, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4, Birgit είπε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7, Sippel, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 1, συμβαστική α, από τέσσερις ομάδες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2, παράγραφος 2, από 4 ομάδες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 11, του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση για την 11 του συντάκτη, άρχεται ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι της ψηφοφορίας. 14 υπέρ, 13 κατά. 8 αποχές. Εγκρίνεται. 12 του συντάκτη πάλι υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3, τροπολογία 13, Τζιν Λάμπερτ, με προφορική τροπολογία. Υπάρχει κάποια αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε τη 13, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 14, παράγραφος 4, ΣΥΠΕΛ, που έχει κάνει και προφορική τροπολογία στην ε, τροπολογία της. με τη 14 και υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 15, Τζιν Λάμπερτ, με προφορική τροπολογία του συγητή. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Ψηφίζεται λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4, η τροπολογία 16, ΣΥΠΕΛ, υπέρ, κατά, αποχές, Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 20 υπέρ. 14 κατά. Εγκρίνεται μεγάλη διαφορά. 17 της υπελπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση. Για τη 17. Ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας. 17 ψήφι υπέρ, 16 κατά, μία, εγκρίνεται, μία αποχή. Παράγραφος 4, τροπολογία 18, Τζιν Λάμπερ, με προφορική τροπολογία του συντάκτη. που είναι η ίδια τροπολογία που κάνει και στην τροπολογία 13. Υπέρ της 18 ως τροποποιήθηκε. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 Τζιν Λάμπερτ πάλι με προφορική τροπολογία του συγητή. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 20, ΣΥΠΕΛ, με κατατμήματα ψηφοφορία, ε, κατόπιν ετήματος των φιλελευθέρων. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ από το without και μετά κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 21, Τζιν Λάμπερτ, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4, τροπολογία 22, Σίπελ με προφορική τροπολογία, δεν υπάρχει αντίρρηση. Ψηφίζουμε λοιπόν υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την 22. Ψήφισαν όλοι, της ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε όλες μαζί τις 23 μέχρι και 31. Ναι ή όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν σύνολο 23, 24 μέχρι και 31 της κυρίας Σίπελ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέραση ψηφοφορία. 33 ψήφοι υπέρ, μία κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στο συντάκτη της γνωμοδότησης. Τα καταφέρατε γιατί όταν ε, το συζητήσαμε δεν φαινόταν τόσο μεγάλη ομοφωνία. Σημείο 8. Τελευταία ψηφοφορία για σήμερα το πρωί. Γνωμοδότηση του Πατρίκ Λεϊαρίκ. Η επί της επιτροπή είναι η Ήτρε για το σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλιβουργία στην Ευρώπη. Παράγραφος 1. Συμβαστική τροπολογία Β. Από πέντε ομάδες υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 36 Δερντέν. υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 28 Σάρια Σεγιά, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 29 Νταρντέν κατά τμήματα από αίτημα των φιλελευθέρων. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα, άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας, 21 υπέρ, 14 κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. Παράγραφος 1, τροπολογία 30, Φρεντερίκ Τερντέν, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία C, παράγραφος 2, από 4 ομάδες υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 36 Νταρντέν, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 38, Σάρια είναι κατά ο εισηγητής, υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση για την 38. Άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας. 16 ψήφοι υπέρ, 17 κατά, 2 αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 2, τροπολογία 39 του Φρεντερίκ Νταρτάιν. Με προφορική τροπολογία, δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, 39 ως τροποποιήθηκε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3, συμβιβαστική D, από τέσσερι ομάδες, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3, 45, Νταρντέν, υπέρ, κατά, αποχές Αν θέλετε να προεδρεύετε εσείς τη θέση σας, μπορείτε κάλλιστα να το κάνετε. Κοιτάξτε αν είστε κατά της απόφασης που λαμβάνω. Λαμβάνω εγώ απόφαση. Επαλήθευση για τις 45. Πέρασε ψηφοφορία 27 ψήφι υπέρ, 8 κατά, καμία αποχή. 47 Εύελιν Ρέγνερ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 46 Στάιρουκ υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρασε της ψηφοφορίας. 18 υπέρ, 17 κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. 48 χάντελ υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. Η 49 είναι παράδεκτη. 50 Κορνέλησεν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 Φρεντερικ Νταρντάν με κατατμήματα ψηφοφορία κατόπιν αιτήματος των φιλελευθέρων. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Για το δεύτερο τμήμα της 51, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. 18 υπέρ, 17 κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. 52 απαράδεκτη, 53 Τόμας Χάντελ υπέρ. Κατά αποχές, επαλήθευση για την 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας, 21 ψήφοι υπέρ, 14 κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. 54 σαριασαγιά με προφορική τροπολογία από τους σοσιαλιστές. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Ο κύριος Οβίρ ενίσταται. Είστε πάνω των τριών αυτοί που είστε αντίθετοι. Ποιος είναι αντίθετος στην προφορική τροπολογία. Πρέπει να είστε τρει. Ποιο είναι αντίθετο στην προφορική τροπολογία. Παρακαλώ. Πολύ ωραία. Εσείς μόνος σας όμως δεν είστε τρία άτομα. Δεν γίνεται δεκτή προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε λοιπόν. Τι συμβαίνει. Αν δεν γίνει δεκτή προφορική τροπολογία, δεν είναι παραδεκτή τροπολογία. Αυτές τις πληροφορίες έχω εγώ. Nous allons travailler en direct ensemble et nous allons Λοιπόν, λοιπόν εργαστούμε μαζί και θα συζητήσουμε κατά πόσο είναι δεκτές κάποιες τροπολογίες. Θα σας διαβάσω την τροπολογία 58 το τμήμα που, θέλετε που μας δημιουργεί πρόβλημα. Θεωρεί, θεωρεί λοιπόν Donc, λοιπόν, θα σας διαβάσω το τμήμα το οποίο πρέπει να ελέγξουμε αν είναι συμβατό με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Απασχόλησης. Θεωρεί ότι οι προτάσεις της Επιτροπής που θέλουν να αντισταθμίσουν την ε, άνοδο της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν καλή πρόθεση, αλλά θεωρεί ότι τα κράτη-μέλη, επειδή αντιμετωπίζουν χρηματοδοτικές δυσχέρειες, και γι' αυτό τον λόγο αυτή η αντιστάθμιση θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο που να εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν το σύστημα <clears throat> ανταλλαγή ε, ποσοστώσεων εκπομπών εξακολουθεί να ισχύει. Συμφωνώ με την άποψη της ελληνική ομάδα. Ή είναι δεκτή αυτή η προφορική τροπολόγηση ή 54 δεν γίνεται παραδεκτή. Τι θέλει το ΕΛΚ. Mondtam, elnök asszony, ezt az utolsó mondatrészt innen, hogy consider the commission... Αυτό το τμήμα θεωρεί ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό το τμήμα θεωρεί ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει να κάνει, ε, τροπολογείται από την προφορική τροπολογία. Αφορά αυτό το τμήμα. Η προφορική που, τροπολογία που λέει ότι θεωρεί ότι η πρόταση Επιτροπής δεν υποστηρίζουμε αυτήν την προφορική τροπολογία. Σας προτείνουμε να ψηφίσουμε χωρίς την προφορική τροπολογία. Πρόεδρος. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Δεν είναι θέμα προφορικής τροπολογίας. Θεωρώ το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 54 εσαγιά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 54 μέχρι εκεί που λέει που οδηγεί στην εξαγω... στις δυνατότητες ε, απασχόλησης και εξαγωγών. Ποιοι είναι υπέρ αυτού του πρώτου τμήματος. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Είναι το κομμάτι που τελειώνει με αποτέλεσμα την εξαγωγή των δυνατοτήτων απασχόλησης. Το ίδιο ισχύει και στι τροπολογίε 55 και 56. Στην παράγραφο 4 ψηφίζουμε τη συμβαστική ε που έχουν υποβάλει 5 ομάδε. Ποιοι είναι υπέρ, αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 4, τροπολογία 64, Νταρντέν, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 4, τροπολογία 65 του Φρεντερίκ Νταρντέν, με προφορική τροπολογία από τη σοσιαλιστική ομάδα. Υπάρχουν αντιρρήσεις σε αυτή την προφορική τροπολογία. Προφορική τροπολόγηση της τροπολογίας. Το ΕΛΚ είναι κατά αυτής της προφορικής τροπολόγησης. Οπότε ψηφίζουμε. δεν έχει να κάνει με το κατά πόσο να αποδεικτεί η τροπολογία 65 ψηφίσμου χωρίς την προφορική τροπολόγηση ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στην παράγραφο 5. Συμβαστική F. Τεσσάρων ομάδων. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 5 έχουμε την τροπολογία 73 με προφορική τροπολόγηση που έχει να κάνει με το αν θα γίνει αποδεκτή. Υπάρχει αντίρρηση στην προφορική τροπολόγηση. Όχι, ωραία, ψηφίζουμε την τροπολογία 73 όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτει. Μετά την παραγραφό 5, τροπολογία 74. Χέντελ, υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. Μετά την παραγραφό 5 πάντα, τροπολογία 75 με προφορική τροπολόγηση. Που ε, έχει να κάνει με το κατά πόσο θα γίνει αποδεκτή αν δεν υπάρχει αντίρρηση στην τροπολόγηση αυτή. Ψηφίζουμε τροπολογία 75 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 76. Νταρντέν με προφορική τροπολόγηση από τους πρασίνους. Υπάρχει αντίρρηση? Όχι. Ψηφίζουμε την 76. Τροποποιηθήσα υπέρ. Κατά αποχές. Να ελέγξουμε την τροπολογία 76. Όπως τροποποιήθηκε από τους πράσινους άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 18 υπέρ, 17 κατά, 0 αποχές πάντα μετά την παράγραφο 5, τροπολογία 77, που θα γίνει αποδεκτή μόνο αν, αν γίνει αποδεκτή η προφορική τροπολόγηση, δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτήν. Ψηφίζουμε την τροπολογία 77 όπως τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. Α, καλά, έλεγχος, Τη 77 σα. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ισοψηφία 16, δύο εποχές. Απορρίπτεται. Μετά την τουλική αναφορά 1, τροπολογία 1 του Νταρδέν, υπέρ κατά εποχές, εγκρίνεται. Πριν, πριν την αιτιολογική σκέψη Α, τροπολογία 2, εισαγιά, αυτή καταπίπτει, ωραία. Οπότε ψηφίσουμε την αιτιολογική Α, στην αιτιολογική Α, τη συμβαστική Α, 4 ομάδων υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται μετά την αιτιολογική σκέψη Α, τροπολογία 7, Νταρντέν υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Μετά την ολική σκέψη α, πάντα τροπολογία 8 ε, του εισηγητή, δύο τμήματα. Ε, ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Α, να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 8 άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 18 υπέρ, 15 κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την λογική σκέψη α, τροπολογία 10, Handel υπέρ, κατά αποχές. Να ελέγξουμε, δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε τη 10, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 29 υπέρ, 0 κατά. Τέσσερις αποχές. Ήταν πεντακάθαρο. Τροπολογία 11. Χωρίς προφορική τροπολόγηση της εν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Νταρντέν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13. Του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15. Χέντελ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17. Νταρντέν υπέρ κατά αποχές. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ και πάλι. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 Νταρντέν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 Νταρντέν υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος. Ελέγχουμε τη 19. Νταρντέν. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 20 υπέρ, 12 κατά. 0 αποχές. Ψηφίζουμε το σύνολο της πρότασης ηλεκτρονικά έρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. είναι υπέρ, 2 κατά, 0 αποχές. Ίδια σχόλια και για τις προηγούμενες εκθέσεις συγχαίρουμε τον εισηγητή μας.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 Chers collègues, alors nous avons Λοιπόν, συνάδελφοι, έχουμε κερδίσει μισή ώρα, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Ελπίζω να μην δημιουργήσει πρόβλημα στη συνέχεια των εργασιών μα. Λοιπόν, όμω αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη σειρά, γιατί η κυρία Όμεν Ρόιτεν που έπρεπε να μιλήσει στο 9 δεν είναι παρούσα. Οπότε θα ασχοληθούμε πρώτα απ' όλα με το 10 που προβλεπόταν ε, για τις 11 και 10. Ελπίζω οι σκιώδεις να μην ενοχληθούν, αλλά εφόσον η συγγήτριά μας ε, Κοστέλο είναι παρούσα, της δίνω το λόγο για να μας πει πώς πήγαν οι εργασίες μας στον τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο για την Ευρωπαϊκή Βοήθεια προς τους απόρους ΦΕΑΝΤ. Ε, κυρία Συγγήτρια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που μπορώ να ενημερώσω την Επιτροπή ότι ο τριμερής διάλογος ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους σκιώδες εισηγητές, το προσωπικό της ομάδας, ε, ε, το προσωπικό και τη γραμματεία του ιδίου του Κοινοβουλίου για την πολύ σκληρή δουλειά που ε, έκαναν για να ολοκληρώσουμε τον τριμερή διάλογο μέχρι την ε, προηγούμενη Πέμπτη. Πολύ δουλειά έγινε, υπήρχαν πολλά τεχνικά κομμάτια τα οποία έπρεπε να ξεκαθαριστούν, αλλά όπως ε, είπα είμαι πολύ ικανοποιημένη που όλα τα θέματα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Στην προηγούμενη συνεδρίαση σας έκανα μια πλήρη επισκόπηση των ε, βασικών θεμάτων που ενδιαφέρουν το Κοινοβούλιο. και χαίρομαι που τα θέματα που ενδιαφέρουν το Κοινοβούλιο ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. 3,5 δις θα είναι ο προϋπολογισμός. Η αρχή της εταιρικής σχέσης που ήταν πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο το να ε, γίνεται διαβούλευση δηλαδή με τις ενδιαφερόμενες ομάδες, ε, να γίνεται παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος, ε, θα συμπεριληφθούν στον κανονισμό και διασφαλίσαμε η αρχή της εταιρικής σχέσης να διασφαλίζεται σε όλο τον κανονισμό. Συνέργειες με πολιτικές που σχετίζονται με τον αγώνα κατά της εσπατάλης τροφίμων, η προώθηση της δημόσιας υγείας, όλα αυτά τα θέματα λύθηκαν με ικανοποιητικό τρόπο. Θα υπάρχουν απλοποιημένες διαδικασίες και αυτό είναι σημαντικό και το Κοινοβούλιο προσπάθησε σε όλα τα στάδια να φροντίσει να μην επιβαρυνθούν ε, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, με διοικητικά καθήκοντα. Ε, καταβάλαμε κάθε προσπάθεια ώστε να έχουμε απλές διαδικασίες. Στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής αναφέρθηκα σε δύο επιχειρησιακά προγράμματα. Θα υπάρχει ένα το οποίο θα έχει να κάνει με την κοινωνική ένταξη των πιο ε, απόρων ε, και θα υπάρχει και άλλο ένα πιο σημαντικό ε, είναι ότι η χρηματοδότηση που είναι μικρή σε σχέση με το σύνολο του προϋπολογισμού αποτελεί όμως σημαντικό ποσό αυτό καθ' αυτό. Σημαντικό λοιπόν είναι η χρηματοδότηση αυτή να χρησιμοποιηθεί ακριβώς για τους πιο άπορους. Αυτή ήταν μια βασική αρχή για το Κοινοβούλιο. Πρόεδρε, όπως γνωρίζουν οι βουλευτές της Επιτροπής μας, Υπάρχουν 40 ε, εκατομμύρια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που, ε, δεν ε, έχουν, που κάθε δύο μέρες δεν έχουν λεφτά για φαΐ. Και είναι τρομακτικό αυτό και χρειάζεται να αναλάβουμε επίγουσα δράση. Το ταμείο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να φτάσουμε τους ανθρώπους αυτούς που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας μας είναι μικρό ταμείο, το αναγνωρίζουμε αυτό, λέμε όμως επίσης ότι το ταμείο αυτό με κανέναν τρόπο δεν αντικαθιστά τις εθνικές πολιτικές για την εφαρμογή των πολιτικών κατά της φτώχειας. Πιστεύουμε ότι το ταμείο αυτό θα αποτελέσει εργαλείο στην καταπολέμηση της φτώχειας γενικά. Να ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι όλους όσους εργάστηκαν σκληρά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα για να διασφαλίσουν Ε, την επιτυχή ολοκλήρωση του τριμερού διαλόγου την προηγούμενη Πέμπτη. Από ό,τι καταλαβαίνω, στις 17 Δεκεμβρίου θα ψηφιστεί στην Επιτροπή το ε, σχετικό έγγραφο και να πω τέλος ότι τα μεταβατικά μέτρα θα ισχύσουν από την αρχή του Δεκεμβρίου, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει διακοπή χρηματοδότησης ε, κανενός ε, από τον οργανισμών ε, και πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Είναι μια εποχή του χρόνου που είναι πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους στους οποίους στοχεύει το πρόγραμμα αυτό και γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρώσουμε το θέμα και να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς στην δύσκολη αυτή περίοδο του χειμώνα. Ευχαριστώ όλους, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς για την ε, βοήθειά σας ε, κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τον τρόπο με τον οποίο ε, χειριστήκατε πολύ σωστά από αρχή μέχρι τέλος, τέλους το θέμα αυτό και συμπεριλάβατε και τις ανησυχίες και άλλων επιτροπών όπως της Επιτροπής Προϋπολογισμών σε τελευταία ανάλυση για το θέμα αυτό νομίζω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να είναι ικανοποιημένο δηλαδή η πλειοψηφία για την υιοθέτηση της εντολής στην Ολομέλεια ήταν σε μεγάλο βαθμό υπέρ της διατήρησης της λογικής, του πνεύματος του προγράμματος. Δηλαδή επιστηστική βοήθεια που να διευρύνεται και με άλλη υλική στήριξη. Και από αυτά που μας είπαν το Συμβούλιο και η Επιτροπή είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη που θα αξιοποιήσουν το δεύτερο τμήμα του προγράμματος για την ε, αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού θα είναι περιορισμένος. Και η κατανομή μεταξύ του προαιρετικού και του υποχρεωτικού τμήματος 2,5 συν 1 δηλαδή, όλα αυτά λοιπόν, στο μεγαλύτερο βαθμό, ακόμη και στο προαιρετικό τμήμα, θα αξιοποιηθούν για το λειτουργικό πρόγραμμα βοήθεια επισητιστική και ηλική στήριξη. Μόνο πέντε χώρε θα ασχοληθούν με το δεύτερο τμήμα όπου θα χρησιμοποιήσουν μόνο το ελάχιστο υποχρεωτικό ποσό. Παρ' όλα αυτά, παρόλα αυτά έχουμε κάποιες ανησυχίες. Είχαμε μάλλον κατά τον τελευταίο τριμερή διάλογο διότι είναι υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μία δήλωση όταν θα εγκριθεί η πρόταση αυτή στην Ολομέλεια. Και θα ζητήσουμε ως συνήθως η Κομισιόν να μας ενημερώσει για το περιεχόμενο αυτής της ανακοίνωσης πριν ανακοινωθεί στην Ολομέλεια για να δούμε αν ε, ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του Κοινοβουλίου, τις ε, προσδοκίες. Δύο σημεία αφορά αυτή η ανακοίνωση. Πρώτον, κάθε πότε θα υποβάλλονται εκθέσεις αποτίμησης και Ποια λογική έχει αυτή η υποχρέωση υποβολής σε σχέση με τις άλλες ε, υποχρεώσεις εκθέσεων στα πλαίσια των πολιτών προοπτικών Αλλιώς, ε, εκτός αν ρυθμιστεί πριν την ψηφοφορία, κατά τεχνικό, το δεύτερο τμήμα που πρέπει οπωσδήποτε να μας ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα κοινωνικά παντοπολία. Όπως φαίνεται, οι διαπραγματευτές μας μας ενημέρωσαν και μετά ξανά άνοιξαν το θέμα αυτό και υπήρχε μια πραγμα... ουσιώδης δυσχέρεια. Διότι το προηγούμενο πρόγραμμα επέτρεπε ε, στα κοινωνικά παντοπολία να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα βοήθεια στους απόρους. Αλλά μετά την έγκριση της ε, νομοθεσίας υπήρξε ένας οριζόντιος κανονισμός της Ένωσης για τα δημοσιονομικά μέσα που απαγόρευε πλέον πλήρως κάθε παρέμβαση μεταξύ ενός προγράμματος του τύπου ταμείου για τους απόρους και τη χρηματοδότηση ενός τμήματος της διανομής βοηθείας. Οπότε, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να δημιουργήσει νέους μηχανισμούς λόγω αυτής της ε, μεταβολής της νομοθεσίας σε ενωσιακό επίπεδο. Για τη χώρα που γνωρίζω καλύτερα, γνωρίζω ότι η γαλλική κυβέρνηση λοιπόν μελετάει μαζί με αυτά τα κοινωνικά παντοπολία πώς θα προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα κατάσταση ούτως ώστε να μπορέσουν ε, τα παντοπολία αυτά να συνεχίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να λειτουργούν. Ωστόσο, επειδή το θέμα αυτό δεν ε, αντιμετωπίζεται εκπεφρασμένα από την νομοθεσία, θέλουμε να δούμε τι δήλωση θα μας κάνει η Κομισιόν κατά την έγκριση του κειμένου. Αυτό ήθελα να αναφέρω. Η κυρία Μωρασουατιέ μου ζητεί στο λόγο και μετά ο κύριος Θέρκας. Μωρασουατιέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την ε, Έμερ Κοστέλο. Η εργασία της ε, ε, ήταν κάτι που περιμέναμε όλοι να δούμε που θα καταλήξει και όλοι ενδιαφερόμασταν πολύ για αυτά. Μας είπατε όμως ότι η Κομισιόν θα μας κάνει τώρα μία δήλωση κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Για αυτήν την δυνατότητα που έχουμε και πάλι για χρηματοδότηση της αγοράς από τα κοινωνικά παντοπολία τροφίμων. Τι θα γίνει στην Ολομέλεια. Θα δούμε συγκεκριμένα τη διατύπωση δηλαδή για να είναι σαφής η κατάσταση ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα δηλαδή ότι όντως υπάρχει σας άκουσα και σας θέτω μια ερώτηση πολύ συγκεκριμένη σας άκουσα κυρία Πρόεδρε σας άκουσα κυρία Πρόεδρε θέτω πολύ συγκεκριμένη ερώτηση και η δεύτερη ερώτηση που θέτω για το θέμα αυτό είναι μήπως επικίνδυνο να αφήσουμε στα κράτη-μέλη τελικά, γιατί από ό,τι κατάλαβα αυτό θα γίνει, να αφήσουμε λοιπόν στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα, εάν και κατά πόσο θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα χρηματοδότησης των ε, κοινωνικών ε, παντοπολίων. Θέρκας και μετά θα απαντήσω. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, σύντομα, να σας πω την άποψη της ομάδος μου. Κάναμε μια συζήτηση για το θέμα αυτό στην ομάδα εργασίας εχθές και οι σοσιαλιστές θέλουν καταρχάς να συγχαρούν δημοσίως την Μερκοστέλο και όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Διότι, κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι αυτή είναι μία από τις σπάνιες στιγμές που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να νιώθει περήφανο, διότι έλυσε προβλήματα ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και αυτό φυσικά έχει στενή σχέση με τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουμε σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι θα περάσουν και τα Χριστούγεννα ευτυχισμένοι και θα μπορούσαν εκατομμύρια από αυτούς να φάνε και να έχουν έστω και το ελάχιστο στο οποίο έχει δικαίωμα ένας άνθρωπος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πέραν από τις λεπτομέρειες, παρά το γεγονός ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα και την ευελιξία και το γεγονός ότι έγιναν σεβαστές κάποιες εθνικές ευαισθησίες, αλλά νομίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι όλοι καταλάβαμε ότι αυτό ε, δεν αφορά μόνο μια χώρα ή κάποιες συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, είναι ένα κοινό πρόβλημα για όλους. Δεν θα πρέπει τα προβλήματα να ε, χωρίζονται αναχώρα, ανα ε, ε, ομάδα, κοινωνική ομάδα. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ταμείο και είναι κοινό το πρόβλημα. Ε, το πρόβλημα είναι κοινό, δεν είναι μόνο για όσους ε, πλήττονται από την απόλυτη ένδια. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή λύση και ότι η Ευρώπη δεν απαντά μόνο στις χρηματοπιστωτικές κρίσεις ή στις κρίσεις των οικονομικών φορέων, αλλά και στις ανθρωπιστικές κρίσεις και στις κρίσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Ε, συγχαρητήρια λοιπόν και στην ΕΜΕΡ και σε όλους τους κοιόδους συζητητές και σε όλους τους συναδέλφους που κατάφεραν να καταλήξουν σε αυτή τη συνένεση και ε, χαίρομαι για το γεγονός ότι η, Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, είχε τον ηγετικό ρόλο σε αυτό το θέμα το τόσο σημαντικό από κοινωνική σκοπιά. Ο Τζαμπόρη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα αντιλαμβάνομαι και το πρόβλημα των κοινωνικών παντοπολίων. Έγιναν διαβουλεύσεις και στη χώρα μου και με αρμόδιες με κυβερνητικές οργανώσεις. Αλλά θεωρώ ότι το πρόβλημα έγκυται αλλού. Δεν έγκυται στο να γνωρίζουμε αν είναι χρήσιμη ή όχι η δραστηριότητά τους. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι είναι χρήσιμα τα κοινωνικά παντοπολία. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην νομοθεσία που έχουμε και αυτή τη στιγμή το ε, κείμενο το οποίο έχουμε εγκρίνει αποκλείει αυτό το ενδεχόμενο. Αντίστοιχα προβλήματα έχουμε αντιμετωπίσει και με άλλες κυβερνητικές οργανώσεις. Υπάρχει ασυμβατότητα ε, με την νομοθεσία. Θα πρέπει να έχουμε παράλληλες δομές, θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των δραστηριοτήτων και έτσι οι οργανώσει που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό θα μπορούν να βρουν και την κατάλληλη λύση. Πρέπει βέβαια να είμαστε και ιδιαίτερα εφευρετικοί σε αυτή την περίπτωση, αλλά δεν χρειάζεται να, να αλλάξουμε εμείς το κείμενο για να βρούμε μια λύση. Υπάρχουν άλλες λύσεις. Πρόκειται για Ε, λύση την οποία θα πρέπει να δεχτούμε. Δεν θα πρέπει να είμαστε κατά τέτοιων λύσεων γιατί είναι πολύ χρήσιμο αυτό που έχουν να προσφέρουν. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Λεαρίκ θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ειλικρινά την κυρία Κοστέλο για τα όσα έκανε και για τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε. Ε, χαιρόμαστε όλοι για το αποτέλεσμα και εσείς κυρία Πρόεδρε και νομίζω ότι ε, καταφέραμε πολλά διότι ε, είναι μια μάχη που δίνουμε εδώ και τρία χρόνια περίπου. για τα κριτήρια τα οποία είχαμε εκφράσει άποψη ευθύ εξ αρχή, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί είμαστε συνολικά ικανοποιημένοι και για τα ποσά και για το γεγονό ότι δεν υπάρχει κάποια διακοπή, διότι θα ξεκινήσει από 1η-1η του 2014 το νέο πρόγραμμα και επομένως ε, θεωρούμε ότι οι αποφάσεις μας έχουν και πολύ σημαντικές συνέπειες ε, για όλες αυτές τις αργωνίες που ασχολούνται με θέματα αλληλεγγύης. Και νομίζω ότι στο γενικότερο κλίμα που έχουμε λίγο πολύ, το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και κατάφερε να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα, είναι αξιοσημείωτο, διότι προσδίδει και πάλι αξία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στους ίδιους ευρωβουλευτές σε ένα πλαίσιο όπου τα θεσμικά όργανα, όπως και εμείς, δεν θα πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις, ε, είμαστε ενώπιον αυτή τη κατάσταση. Βεβαίω δεν ήταν καλύτερα να μην έχουμε απόρους, αλλά είναι και καλό το αποτέλεσμα που έχουμε. Κύριε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι γενικά μπορούμε να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα ε, αυτού του θέματος. Ε, ήταν επίμαχο θέμα εντός του Κοινοβουλίου, εντός του Συμβουλίου, μεταξύ ημών και του Συμβουλίου. Ε, νομίζω Πάντως ότι η κυρία Κοστέλο και η Πρόεδρος έκαναν, ε, τα καταφέραν πολύ καλά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ε, φαίνεται ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι με τα ποσά που θα λάβουν και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε περήφανοι που βελτιώσαμε τις ε, δυνατότητες για τις ε, οργανώσεις βοήθειας να χρησιμοποιούν τα ε, χρήματα εκεί που τα χρειάζονται περισσότερο. Κυρίως θα πρόκειται για παροχή τροφίμων, μπορεί όμως ε, και να είναι πράγματα όπως προγράμματα ή τρόποι αποφυγής σπατάλης των τροφίμων. Και υπάρχουν επίσης μέτρα κοινωνικής ένταξης για να βοηθηθούν οι πιο στερημένοι. Γενικά, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, θα δώσω το λόγο και στην εισηγήτρια, αλλά ευχαριστώ που αναφέρατε το σημείο, το είχε αναφέρει η εισηγήτρια, η καταπολέμηση της πατάλης τροφίμων. Και όπως και η εισηγήτρια, έχουμε επιμείνει το λειτουργικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αποκλεισμών να μην είναι αντιγραφή του κοινωνικού ταμείου. Ναι, μεν υπάρχει μια ασάφεια για τον όρο. Για αυτά τα παντοπολία. Μα νομίζω ότι είπα σαφώ ότι δεν έχει ανοίξει η πόρτα. Έχει κλείσει η πόρτα. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα τα κοινωνικά παντοπολία να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό που ζητήσαμε από την Επιτροπή είναι να κάνει μια δήλωση στην οποία θα πει συγκεκριμένα τους λόγους για τους οποίους αρνήθηκε να ξανανοίξει αυτή η πόρτα. Οπότε επανερχόμεθα όπως ε, το είπε σαφώς και ο Τσαουρί σε ευθύνη των κρατών μελών. Και για τη χώρα όπου, από όπου προερχόμεθα και η κυρία Μωρά και εγώ έχουμε ήδη απευθυνθεί στην κυβέρνηση και τις έχουμε ζητήσει να κάνει ό,τι χρειάζεται για να μπορέσουν να συνεχίσουν να βοηθούν τους πιο στερημένους, τους πιο απόρους, επικοδομητικά αυτά τα παντοπολία. Απολογισμός του προγράμματος αυτού. Ευχαριστώ τον κύριο Λουγκαρίκη για αυτά που είπε, γιατί έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο. Εμείς ήμασταν αυτοί που επιμείναμε για αυτό το πρόγραμμα να θυμάστε ότι όταν εγκρίθηκε στην Ολομέλεια το θέμα αυτό, νομίζω πως ήταν το Φεβρουάριο του 2012, μέσω ενός ψηφίσματος που επέμενε ότι πρέπει να διατηρηθεί αυτό το πρόγραμμα. Τότε το Συμβούλιο ήθελε να το καταργήσει. Και τότε, αλλά και μετά, χρειάστηκε να συνεχίσουμε, να επιμείνουμε για να συνεχιστεί το 2013 και το 14 το πρόγραμμα αυτό, γιατί ορισμένοι ήθελαν να το καταργήσουν. Γι' αυτό επειδή επιμείναμε και επειδή άλλαξε και η κατάσταση στο Συμβούλιο, γι' αυτό παραμένει αυτό το πρόγραμμα, έχει γίνει υποχρεωτικό και γι' αυτό έχει και επαρκεί ή τουλάχιστον αυτή την χρηματοδότηση. Νομίζω ότι υπάρχει λοιπόν μια συμβολή του Κοινοβουλίου η οποία πρέπει να επενεθεί και για την οποία ευχαριστούμε πολύ την συγκήτριά μας. Κυρία Κοστέλο θέλετε να επανέλθετε ή όχι. Α παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και, και ευχαριστώ όλους ε, για τις παρατηρήσεις τους. Ε, τα περισσότερα θέματα έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα, αλλά θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι το πρόγραμμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θα πρέπει να θεωρηθεί ε, και πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το προηγούμενο πρόγραμμα προερχόταν ε, από τον ε, προϋπολογισμό της Γεωργίας και δεν θεωρήθηκε κοινωνικό μέτρο. Τώρα όμως μιλάμε για τους ανθρώπους που είναι άποροι, που δεν έχουν να φάνε. Αλλά και οι οργανώσεις που μοιράζουν τρόφιμα ε, επίσης ε, παρέχουν μέτρα κοινωνικής ένταξης ε, και είναι σημαντικό ότι το θέμα αυτό πλέον θεωρείται θέμα κοινωνικών υποθέσεων. Η κοινωνική ένταξη αποτελεί κεντρική, κεντρικό ενδιαφέρον των οργανώσεων που παρέχουν τα τρόφιμα. Τα τρόφιμα φυσικά είναι πολύ σημαντικά. Ε, και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λαμβάνουν πακέτα τροφίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ όλους ε, τους ε, συναδέρφους που αναφέρθηκαν στο θέμα της πατάλης των τροφίμων, την πρόθεση υγιεινή τρόπου ζωής, το μοίρασμα των πακέτων τροφίμων κλπ. Νομίζω ότι έχουμε βελτιώσει την πρόταση της Κομισιόν στα θέματα αυτά. Επίσης έχουμε ένα καλό πρόγραμμα για τη ε, διάδοση των αποτελεσμάτων ε, και πλατφόρμα για ε, την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. Δεν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με τον ε, ρόλο των, ε, μικρο... των μη κυβερνητικών ε, οργανώσεων και των άλλων φορέων που συμμετέχουν σε αυτά. Έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Συζήτησαν μεταξύ του το, το... το πρόγραμμα αυτό, συνομίλησαν και μαζί μα και ελπίζω ότι είναι και αυτοί ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα που έχουμε μπροστά μα. Όσον αφορά τα κοινωνικά παντοπολία, Πρόεδρε, νομίζω ότι το αναφέρατε κι εσείς. Είναι ένα θέμα που επαναφέραμε στις διαπραγματεύσεις, αγωνιστήκαμε. Μπορεί τελικά να μην είχαμε το αποτέλεσμα που προτιμούσαμε, ελπίζουμε όμως ε, οι χώρες να μπορέσουν ε, να δημιουργήσουν τέτοια παντοπολία στα κράτη-μέλη παρόλα αυτά. Ε, ευχαριστώ λοιπόν θερμά όλους. Ευχαριστώ το προσωπικό του Κοινοβουλίου, το προσωπικό της Κομισιόν, ε, τις πολιτικές ομάδες ε, και όλους όσους ξενύχθησαν προσπαθώντας ε, να λύσουν τις κρεμότητες που είχαμε. Νομίζω ότι η πρόταση τελικά που έχουμε είναι πολύ καλή. Très bien. Alors, nous en venons à un dossier. Ωραία. Περνάμε σε ένα ακόμα θέμα το οποίο στέφθηκε με επιτυχία. Σημείο 9. Διαπραγματεύσεις με τη Συμβούλιο σχετικά με τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Μπορεί βέβαια να αφορά λίγο λιγότερους, αλλά και πάλι είναι κοινωνικό ζήτημα. Αποτελέσματα λοιπόν του τελευταίου τριμερούς διαλόγου με την Λιθουανική Προεδρία για μια έκθεση για την οποία ήταν αρμόδια η κυρία Όμενε Ρόιτερ. Της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους εργάστηκαν πάνω στο θέμα αυτό και μας βοηθήσαν να πετύχουμε ε, τόσο καλό αποτέλεσμα. Είμαι ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα. Στην αρχή είχαμε ένα σχέδιο οδηγίας ε, το οποίο υποπλήθηκε από την Κομισιόν μας είπε η Κομισιόν ότι ο κόσμος εξοικονομεί, ε, αποταμιεύει χρήματα σε κάποιο ε, ε, συνταξιδοτικό ταμείο, θέλει να τα μεταφέρει σε άλλο. Διαπιστώσαμε πολύ σύντομα ότι η μεταφορά κεφαλαίων ήταν πολύ δύσκολη, ακόμα και σε χώρες όπου ήδη γινόταν. Συνεχίζει να γίνεται αυτό στις κάτω χώρες, αλλά είναι πολύ δύσκολη η μεταφορά των χρημάτων. Είπαμε λοιπόν και εμείς στο Κοινοβούλιο ότι θα είναι καλύτερο να εξετάσουμε το δικαίωμα μεταφοράς και μήπως ε, μπορεί να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς ε, των ε, δικαιωμάτων και δεδομένου του τρόπου που λειτουργούν οι συμπληρωματικές συντάξεις. Υπάρχουν κάποια κρατημέλη που έχουν τέτοια τέτοια υπάρχουν όμως άλλα κρατημέλη που έχουν οργανώσει με τελείως διαφορετικό τρόπο τα στεξιδοτικά τους ταμεία. Θέλουμε να αποφύγουμε, να αρχίσουμε να παρεμβαίνουμε στον τρόπο που τα κράτη-μέλη οργανώνουν τα, ταμεία, τα συνταξιδοτικά ταμεία. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε όμως είναι να διευκολύνουμε την κινητικότητα, την ελεύθερη κινητικότητα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει εργαστεί κάπου, να έχει τη δυνατότητα όχι να τιμωρείται αν εργαστεί για άλλον εργοδότη ή μετακομίσει σε ξένη χώρα. αλλά να ανταμείβεται γι' αυτό. Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα για την κινητικότητα στην Ευρώπη. Αυτό είναι σημαντικό. Μετά από, αντίδραση, μετά από την απάντηση του Κοινοβουλίου και ε, ε, κάποιες παρατηρήσεις από την Κομισιόν, το θέμα αυτό πήγε στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο είπε ότι είναι σημαντική κινητικότητα. Θέλουμε όμως να φροντίσουμε να υπάρχει πλεονέκτημα ε, μόνο εάν ε, μετακομίσει κανείς σε ξένη χώρα, το οποίο σημαίνει ότι η πρόταση αυτή εξετάζει τα ελάχιστα πρότυπα για ε, απόκτηση και πληρωμή σύνταξης σε περίπτωση που κάποιος μετακομίζει σε ξένη χώρα, σε άλλο κράτος μέλος και έχουν αποκλείσει από το πεδίο εφαρμογή ε, την ε, μετακίνηση εντός του ιδίου κράτους μέλους. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα ε, κάποια προβλήματα και οι εργαζόμενοι που μετακομίζουν από, μία, από ένα κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος έχουν καλύτερες προϋποθέσεις από αυτούς που μετακομίζουν εντός του ιδίου κράτους μέλους. Δεχτήκαμε την πρόταση αυτή. Τα ίδια τα κράτη-μέλη μας έδωσαν ε, αιτιολόγηση. Μας είπαν ότι στο χρόνο που απομένει για την εφαρμογή αυτού του μέτρου ε, και μέχρι τη θέση σε ισχύ θα ε, βελτιώσουν τις προϋποθέσεις εντός των χωρών τους. Δεν ήταν πολύ εύκολο το δεχτούμε αυτό, αλλά αν δεν το δεχόμασταν δεν θα είχαμε καθόλου σχετική οδηγία. Επίσης αναφέρθηκαν κάποια πρότυπα για, την, ε, ε, για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Σε κάποιες χώρες ε, ξεκινάει κανείς να εξασφαλίζει συνταξιοδοτικά δικαιώματα στην ηλικία των 21 ετών. Στη Γερμανία, στο Λουξεμβούργο η τάση είναι να είναι κανείς μεγαλύτερο στην ηλικία. Στη Γερμανία περίπου 25 χρόνια. Και χρειάζεται 20, χρειάζονται 25 χρόνια, το οποίο σημαίνει ότι ε, αν ε, ε, κάποιος είναι, ξεκινήσει να δουλεύει σε ηλικία 29,5 ετών μετά από, και μετά αλλάξει εργοδότη, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει συνταξιδιωτικά δικαιώματα. Είπανε λοιπόν οι, τα κράτη-μέλη ότι θα βελτιώσουν την κατάσταση εντός των χωρών τους. στην νομοθεσία αυτή ε, μιλάμε για μια περίοδο εξασφάλισης ταξιδιωτικών δικαιωμάτων που ξεκινάει από την ηλικία των 21 ετών. και υπάρχει ε, έτος ε, αναμονής τουλάχιστον τριών ετών, το οποίο αποτελεί σαφή βελτίωση σε σχέση με την κατάσταση που είχαμε πριν από όλα αυτά. Και έπρεπε να αγωνιστούμε σκληρά για να περάσουν οι θέσεις μας, αλλά Νομίζω ότι η προϋπόθεση αυτή που θέσαμε βελτιώνει τις προϋποθέσεις για την ελεύθερη κινητικότητα. Αυτό που θέλαμε να πετύχουμε ήταν το εξής. Θέλαμε να αποφύγουμε ο κόσμος ε, να ε, έχει εξασφαλίσει ταξιδιωτικά δικαιώματα ε, μέσα σε τρία χρόνια και να πληρώνεται αμέσως το κεφάλαιο, γιατί αυτό σημαίνει ότι όταν φτάσει κανείς στην ηλικία συνταξιοδότησης δεν θα έχει πια δικαίωμα σε σύνταξη. Και αυτό ήταν θέμα που συζητήθηκε μέχρι το τέλος. Και αν μιλάμε για μικρό ποσό, τότε οι συνεισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών μπορούν να πληρωθούν αλλά το πρόσωπο που θα λαμβάνει τις πληρωμές αυτές θα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του να, ή να έχει την επιλογή να γίνει η πληρωμή ή να διατηρήσει ε, τα συνταξιδοτικά δικαιώματα. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, ε, λοιπόν, ε, ε, εξετάζουμε την ε, περίοδο θέσης ε, σε ισχύ. 3 συν 2 ήταν αρχικά αυτό που θέλαμε. Τώρα εξετάζουμε περίοδο μεταβατική 4 ετών. Τα τρία χρόνια ήταν για όλους. Τα δύο επιπλέον έτη ήταν για τις περιπτώσεις όπου υπήρχαν προβλήματα. Και πρόεδρε, τώρα έχουμε τέσσερα χρόνια για όλους και το δεχτήκαμε αυτό. Νομίζω ότι κάλυψα όλες τις πτυχές του θέματος αυτού. Αυτά ήταν τα σημεία που θεωρήσαμε εμείς σημαντικά. Πρόκειται για μια πρόταση με την οποία πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε απολύτω ε, ικανοποιημένοι, διότι βελτιώνει την ελεύθερη κινητικότητα των ε, ανθρώπων και θα λειτουργεί καλύτερη η ελεύθερη κινητικότητα από το και Ευχαριστώ, Ποιο θέλει το λόγο μετά, ο Μαν. Και αυτά είναι όλα. Ο κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι μάλλον λακωνικός, διότι η Ρία μας εξήγησε πολύ καλά τα διάφορα ε, σημεία στα οποία είχαμε επιτυχία και τη συγχαίρω και για τα όσα έκανα αυτή και για όσα κάνετε και εσείς κυρία Πρόεδρε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων καταφέραμε να έχουμε πραγματική πρόοδο και να έχουμε πραγματική δυνατότητα μεταφοράς ε, και κάτι το οποίο ευνοεί την ελεύθερη κυκλοφορία και φυσικά είναι και υπέρ του εργαζομένου ε, για τη μελλοντική του ε, συνταξιοδότηση όποτε τη χρειαστεί. Είμαι πολύ ικανοποιημένος λοιπόν από το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης. Ο Τόμας Μάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και και τους άλλους γιατί δεν ήταν εύκολο να επιτύχει κανείς συμβασμούς αν θέλει να έχει κάποιο επίπεδο. Και στην Γερμανία θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε κάποιο επίπεδο. Αλλά χρειαζόμαστε κοινέ λύσεις για να μην έχουμε κινητικότητα ε, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στις πράξεις. Ο συμβασμός με τα... για την ηλικία 21 ε, ετών και την περίοδο αναμονής 3 ετών εντάξει είναι κάπως επίπονο αλλά σε τελευταία ανάλυση Εφόσον καταφέραμε να συμφωνήσουμε και οι τρεις, ε, αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα. Ελπίζω όμως ε, να μην ξαναζητηθεί το θέμα αυτό και ε, να μην υπάρξουν νέες ρυθμίσει σε δύο-τρία χρόνια. Πρέπει να υπάρχει σταθερότητα για το θέμα αυτό. Και νομίζω ότι έχουμε μια καλή βάση για να υπάρξει σταθερότητα, για να ενημερώσουμε. Γιατί εμείς που ασχοληθήκαμε τόσα χρόνια με το θέμα αυτό έχουμε ευθύνη να ενημερώσουμε για το τι επιτύχαμε. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ, θεωρώ ότι ήταν καλό. Ε, το ότι επίσης είπαμε ότι ε, για ορισμένα θέματα ε, δεν, έχουν προχωρήσει, δεν έχουμε προχωρήσει όπως θέλαμε, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει σταθερότητα, να διατηρηθεί σταθερό αυτό το πλαίσιο, θα ήταν σημαντικό πολιτικό μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής που δέχτηκαν να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις χωρίς να ξαναδούμε την εντολή που είχε δοθεί κατά την προηγούμενη θητεία στην κυρία Ομαν Ρόιτεν. Αυτό μας, επιτρέπει, μας επέτρεψε να κλείσουμε το θέμα κατά την ε, παρούσα θητεία χωρίς αναδιαπραγμάτευση. Υπογραμμίζω ότι ενωμένα ενήργησε η διαπραγματευτική μας ομάδα ούτως ώστε αυτή η οδηγία να μην παίξει μόνο το ρόλο τα πιο λαμπρά στοιχεία να μπορούν να ε, κινηθούν από ένα μέρος στο άλλο αλλά θα πρέπει ε, φυσικά και οι συνταξιούχοι να μπορέσουν να έχουν δυνατότητα στην ελεύθερη διακίνηση με μεταφορά των δικαιωμάτων τους, των συνταξιδοτικών, με την συνένεσή τους. Εάν δηλαδή, δηλαδή από τη στιγμή που θα γίνουν απαιτητά τα δικαιώματά τους θα είναι δυνατόν να τα αξιοποιήσουν. Να υπάρχει όμως και η συνένεση του εργαζομένου για έναν τέτοιο μηχανισμό. Σημειώνω ωστόσο ότι η αντιμετώπιση του Συμβουλίου ήταν πολύ διαφορετική. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν με πολύ άτυπο και ελαφρό τρόπο τα κράτη-μέλη να επιτρέψουν δηλαδή στους εργαζομένους, στους μισθωτούς των χωρών τους ένα παρόμοιο καθεστώς ε, δυνατότητας μεταφοράς, φοβάμαι ότι αυτές οι δεσμεύσεις είναι κάπως προαιρετικές. Άρα μπορεί να εισάγουμε διακρίσεις στην ουσία μεταξύ των ε, εργαζομένων που μπορούν να μεταφέρουν αυτά τα δικαιώματα όταν πηγαίνουν από μια χώρα στην άλλη και εκείνων που μετακινούνται εντός μιας χώρας. Νομίζω ότι η διαδοχή μας θα πρέπει να ξαναδούν το θέμα αυτό Άρα ε, δεν κλείνουμε πλήρω το θέμα αυτό. Κυρία Συγήτρια, θέλετε να προσθέσετε τίποτα. Νομίζω ότι υπόθηκαν όλα. Νομίζω ότι πολλοί συνέβαλαν ε, στην επίτευξη αυτής της ε, συμφωνίας. Και η Κομισιόν κατέλαβε σημαντικές προσπάθειες ε, για, να μπορέσει να υποβάλει συμβαστικές προτάσεις και θα ήθελα να του ευχαριστήσω γι' αυτό. Ε, είχα ε, ανταλλαγή email, κάποιοι ευρωβουλευτές ε, είχαν ανταλλαγή email με τους, με την ε, γερμανική μια αντιπροσωπεία. Ε, μάλλον έγινε ανταλλαγή ε, email, στην οποία όμως δεν συμμετείχε η συγγήτρια. κυρία Πρόεδρε, δεν θα έπρεπε να εργαζόμαστε έτσι. πιστεύω ότι θα ήταν καλό να το συζητήσουμε αυτό λίγο. Άλλες μόνιμες αντιπροσωπείες κρατών μελών κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω θερμά γι' αυτό. Ξέρουν ε, οι χώρες αυτές ε, ε, ότι μιλάω για αυτές. Χάρη λοιπόν στην, στην συλλογική προσπάθεια πετύχαμε τόσα πολλά. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον Φρεντερίκ. συνεργαστήκαμε πολύ καλά και αν υπάρχει εμπιστοσύνη, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Στην ανταλλαγή email που είχαμε, Ε, νομίζω δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς την εισηγήτρια ότι δεν έκανε τη δουλειά της. Ε, τα αποτελέσματα αυτά λοιπόν ε, είναι αποτελέσματα της καλής μας συνεργασίας. Ευχαριστώ και σένα, Τζιν. Ευχαριστώ. Η διαδικασία είναι κάπως ασυνήθιστη σε σχέση με τη συνήθη πρακτική μας. Πρόκειται για δεύτερη ανάγνωση. Θα ψηφίσουμε λοιπόν τη θέση της Επιτροπής ε, Απασχόλησης ε, που είναι σύμφωνη με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στις 9 Δεκεμβρίου και μετά θα γράψω ένα επίσημο γράμμα στο Συμβούλιο που μετά από, την, ε, από τον έλεγχο του κειμένου από τους ε, ε, γλωσσομαθείς νομικούς λοιπά, θα μας στείλει γύρω στα μέσα Φεβρουαρίου την θέση του Συμβουλίου που θα μας επιτρέπει να εγκρίνουμε το σχέδιο σύσταση στη δεύτερη ανάγνωση και να περάσουμε τον Απρίλιο στην Ολομέλεια. Αυτό το θέμα λοιπόν θα μας απασχολήσει μέχρι το τέλος της θητείας όταν ανέλαβα την Προεδρία, μεταξύ των θεμάτων που ήταν ε, υποεξέταση, ήδη υπήρχε. Οπότε, να περάσω στο επόμενο θέμα, το 11, όπου δίνω το λόγο για τις ε, πτυχές απασχόληση και κοινωνικά θέματα της ετήσιας επισκόπησης ανάπτυξης στον εισηγητή μας Σέρχιο Ουτιέρες Πριέτο θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής του. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι η τρίτη έκθεση που κάνουμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και η δεύτερη που κάνουμε ευτυχώς στο ίδιο επίπεδο που έκανε και η ΕΚΟΝ. Αυτό σημαίνει τη σημασία έχουν τα κοινωνικά θέματα, κυρίως η απασχόληση και ο μακροοικονομικός συντονισμός, συντονισμός της λεγόμενης διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Καταρχάς, να κάνω μια δήλωση ε, προθέσεων που δεν είναι αυτονόητη αλλά σημαντική. Η σημαντική είναι η προσπάθεια διαλόγου και συνένεσης. Πρέπει να ανταλλάξουμε απόψεις για την πραγματικότητα όπως τη ζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή που οι ανισότητες αυξάνονται αλλά και οι αποκλίσεις ε, μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Μιλάω για ανισότητες ε, γεωγραφικές. Χρειάζεται λοιπόν συνένεση. Γιατί νομίζω ότι για να επιτύχουμε το καλύτερο πριν τα κράτη-μέλη κάνουν τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων είναι να στείλουμε λοιπόν σαφή μηνύματα προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή για συγκεκριμένα θέματα που τα συζητάμε σε κάθε έκθεση που μας απασχολεί και που το θέμα δεν είναι μόνο να είναι σε εκθέσεις μας αλλά να μπουν και στις πολιτικές που θα μπουν στις πολιτικές, μετα... στις πολιτικές μεταρρυθμίσεων των διαφόρων κρατών μελών. Τι θέλουμε να κάνουμε αυτή την έκθεση. Το πρώτο, το πρώτο απ' όλο είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός από πλευράς της Επιτροπής ε, Απασχόληση. Βεβαίως η Κομισιόν προσπαθεί να υπογραμμίσει τα θετικά στοιχεία κυρίως μακροοικονομικά που βοηθάνε την ανάκαμψη. Αλλά σημαντικό είναι ότι εμείς ως Επιτροπή είναι να συνεχίζουμε να τονίζουμε ότι συνεχίζουν να χάνονται θέσεις εργασίας, ότι οι νέοι θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό στην ε, ανεργία, αυξάνεται ο κοινωνικός αποκλεισμό, αυξάνεται η φτώχεια. Τα κράτη-μέλη λοιπόν πρέπει να έχουν μια πολύ ισχυρή πολιτική για να, για να αλλάξει ριζικά η τάση για τα θέματα αυτά, που είναι η δική μας αρμοδιότητα εδώ. Το πιο σημαντικό είναι λοιπόν να μην υπάρξει εφησυχασμός. Υπάρχει ακόμη και συνεχίζεται μια κοινωνική κρίση που δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να αντιμετωπίσουμε. Και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε περισσότερα στοιχεία. Πρέπει να υπογραμμίσουμε λοιπόν τα πιο σημαντικά θέματα για μας. Θέλουμε να ενισχύσουμε λοιπόν κάποιες απόψεις που ήδη έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες εκθέσεις. Πρώτον, σημασία των κοινωνικών δικτών. Είναι κάτι καινούριο που έχουμε σε αυτή τη διαδικασία του εξαμήνου που ξεκινάει τώρα. Αλλά δεν είναι ούτε επαρκείς ούτε υποχρεωτικές, όπως ακριβώς είχαμε απαιτήσει ως Επιτροπή. Θα έπρεπε οι κοινωνικές πτυχές να αναλύονται όπως και οι, να αναλύονται όπως και οι μακροοικονομικές πλευρές γιατί τα κοινωνικά θέματα παίζουν μεγάλο ρόλο Επίσης θέλουμε να δημιουργηθεί ένα Eurogroup για κοινωνικά θέματα και απασχόλησης για να τονίσουμε την ισότιμη σημασία που πρέπει να έχουν αυτές οι πολιτικές και τώρα και για το μέλλον. Βεβαίως, η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας παραγωγικότητας πρέπει να βασίζεται από τη μία στις επενδύσεις στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Δεύτερη, δεύτερος πυλώνας της προσπάθειας πρέπει να είναι η εκπαίδευση. Το συζητήσαμε και χθε όπου είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε ακόμη μεγάλες προσπάθειες στον τομέα αυτό δεν θα πρέπει δηλαδή η δημοσιονομική εξυγίανση να περιορίζει της εκπαίδευση. Και το τρίτο, ο τρίτος πυλώνας πρέπει να είναι η καινοτομία. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, αλλά όχι οποιασδήποτε θέσεις εργασίας. Αυτό είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, που το βάλαμε και στην έκθεση Λόπε Φοντανέ και της κυρίας Μπερές στα προηγούμενα εξάμεινα. Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της ε, αγοράς εργασίας πρέπει να συνδυάζει πολύ ε, ορθά την ασφάλεια με την ευελιξία. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τη φτώχεια στην Ήπειρό μας και συνεχίζουμε να προειδοποιούμε ότι είναι αναγκαίο να ενταθούν οι προσπάθειες και της Ένωσης και των κρατών μελών για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Κατά την ε, ενδιάμεση αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να κάνουμε όλες τις αναγκαίες επαληθεύσεις για να δούμε αν τα 7 δις που έχουμε αφιερώσει σε αυτό το στόχο είναι επαρκή ή αν θα πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση αυτής της προσπάθειας όπως ζήτησε η Επιτροπή μας και όπως ε, απαιτεί και ο διεθνής, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Τονίζουμε επίσης το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια καλύτερα, Έχουμε ασχοληθεί πολύ με το δημόσιο χρέος και φυσικά πρέπει να συνεχίσουμε να ασχολούμεθα με αυτό το δημόσιο χρέος, αλλά υπάρχει και πρόβλημα ιδιωτικού χρέους που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν σχέδια αναδιάρθρωσης και αυτού του χρέους. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν προγράμματα για χρηματοδότηση των μικρομεσαίων αλλά και των οικογενειών είναι σημαντικό στοιχείο αυτό για έξοδο από την κρίση και για να επανέλθουμε στην οικονομική ανάπτυξη. Νομίζουμε λοιπόν ότι η έκθεση είναι πολύ οριζόντια, ασχολείται με τα σημεία κλειδιά που πρέπει να τονίσει η Επιτροπή Απασχόλησης Κοινωνικών Θεμάτων. Είναι λοιπόν σημαντική η προσπάθεια διαλόγου και εξέβρεσης συνένεσης για να καρποφορήσουν οι προσπάθειές μας που θα καταλήξουν στα, σχετικά, στα εθνικά σχέδια μεταρρυθμίσεων. Ευχαριστώ πολύ. η Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ και η Μαρίς Κορνέλισεν, αλλά πριν από αυτό να κάνω μια παρατήρηση, γιατί νομίζω ότι όλα όσα μας προτείνει ο εισηγητής μας είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να μας απασχολήσουν ιδιαίτερα εδώ στην Επιτροπή μας. Εγώ όμως, ως πρόεδρος επιτροπής μας, έχω την εξή ανησυχία. Θέλω να είναι ρεαλιστικά αυτά που κάνουμε και να περάσουμε από το τοπικό στο πραγματικό. Και η πραγματικότητα είναι η αντιπαράθεση που έχουμε να κάνουμε με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Και το εφαλτήριο της συζήτησής μας εδώ θα πρέπει να είναι το η ετήσια έκθεση ανάπτυξης όπως μας την έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει Πρέπει να έχει βάση την ετήσια έκθεση ανάπτυξης, να δούμε τι έχουμε και από εκεί και πέρα να τη συμπληρώσουμε. Εμείς όμως θα, θα μπορούσαμε να τα ξαναγράψουμε όλα για να ευχαριστηθούμε και να εκνευρίσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ε, δεν μπορούμε να ξεκινούμε από αυτή τη θέση ε, δεδομένου ότι έχουμε μια λογική συναπόφαση που είναι η μόνιμη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, της Επιτροπής μας αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να έχουμε συναπόφαση και νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε τις προτάσεις μας και ε, να δούμε και τι πρέπει να τροποποιήσουμε στην ετήσια έκτηση ανάπτυξης. Ε, είναι πολύ πλούσια η έκθεση και στον τό χρόνο ρεκόρ που μας έχει δοθεί θα πρέπει να δούμε με τις τροπολογίες μας πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Η Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ, η κυρία Κορνέλεσον, η κυρία Χάρκινγκ, η Έντιτ Μπάουερ και αυτές νομίζω ήταν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, νομίζω ότι το πρώτο θέμα θα μπορούσε να ήταν η διαμαρτυρία για τον ελάχιστο χρόνο που μας δίνεται η έκθεση ούτε καν είχε μεταφραστεί, έπρεπε να εργαστούμε στα αγγλικά και έχουμε και μια προθεσμία κατάθεση τροπολογιών μέχρι την Τρίτη. Δυστυχώς, αν το συγκρίνουμε αυτό με τις προθεσμίες που έχει ε, η Επιτροπή ε, η αρμόδια, η οποία έχει πολύ περισσότερο χρόνο στη διάθεσή της και έχει και όλες και τις διακοπές των Χριστουγέννων για να καταθέσει τροπολογίες. Είναι πολύ πλούσια η έκθεση του Σέρχιο και είναι πολύ δύσκολο να τη συζητήσουμε όλα ε, την έκθεση μία προς μία. Να πω απλώς ότι εμείς από πλευράς ΕΛΚ είμαστε θετικοί σε οποιαδήποτε συμφωνία, αλλά βεβαίως υπάρχουν και κάποια σημεία τα οποία θα υπάρχουν διάσταση απόψεων και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να τα εξηγήσω. Πρώτον, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία ε, με βρίσκουν σύμφωνοι. Ε, μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο επικεντρώνεται ο κύριος Γκουτιέρες, ε, επικεντρώνεται στη δημοκρατική ε, συμμετοχή, τη σχέση με την ένδια και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αύξηση του προπολογισμού για πρωτοβουλίες για την ε, ε, ανεργία των νέων και για όλα τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τη φτώχεια, την μακράς διάρκεια ανεργίας, προβλήματα γυναικών και άλλων υπολείπων ευπαθών ομάδων και όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάζουμε και να προτείνουμε λύσεις και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να υπάρχουν οι βέλτιστε δυνατές λύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ διαφωνώ λίγο με την Πρόεδρο και θεωρώ ότι το σχέδιο έκθεσης που μας έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα τα οποία πρέπει ακόμα να επεξεργαστούμε, τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, να ευνοήσουμε τη δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι πολύ σημαντικό και να δούμε πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο με τον κύριο Κουτιέρες, κυρίως ε, όλα τα θέματα που αφορούν ε, την ε, δημοσιονομική εξυγίανση. για την ομάδα μας το θέμα της δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι πολύ σημαντικό διότι αποφέρει καρπούς και αυτό το βλέπουμε με αυτά αποτελέσματα στην Ισπανία. Εκεί που είχαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, άρχισαν να βελτιώνονται τα πράγματα και θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα θέλουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα και μας το είπαν και οι Επίτροποι προχθές, ο κύριος Σάντορ, και το πώς βελτιώθηκε η κατάσταση χάρη στις προσπάθειες οι οποίες κατεβλήθησαν και τώρα πλέον μπορεί να δοθεί μεγαλύτερο περιθώριο για πολιτικές ανάπτυξης και απασχόλησης. Βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται και με την κατάλληλη εξυγίανση για να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη. Και νομίζω ότι αυτή θα είναι η τοποθέτηση του ΕΛΚ, όπως είπαμε και στην προηγούμενη ε, έκθεση. Ναι μεν δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά με τη δέους ευελιξία. Υπάρχει στην έκθεση του κυρίου Γκουτιέρεθ ε, μια σειρά από επικρίσεις ή τουλάχιστον έτσι τις ερμηνεύω εγώ για τις πολιτικές των τελευταίων δύο-τριών ετών και δεν συμφωνώ με αυτές τις επικρίσεις διότι θεωρώ ότι αποφέρουν καρπούς. Ε, τίποτα άλλο. Να πω ότι προσβλέπω σε μια στενή συνεργασία για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια έκθεση στην οποία θα υπάρχει ευρεία συνένεση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κορνέλησεν και μετά η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τον εισηγητή, συγγνώμη, για ένα πολύ καλό σχέδιο κειμένου. Οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι λίγο θλιβερό το γεγονός ότι μοιάζει πολύ με τις εκθέσεις που έκανα εγώ το 2012 και τις εκθέσεις που έκανε η κυρία Λόπε Φοντανιέ στις αρχές του έτους το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ό,τι φαίνεται μας αγνοούν παντελώς κάθε χρόνο και ίσως καλό θα ήταν να εξετάσουμε λίγο προσεκτικά ε, ότερα τη διαδικασία. Έχουμε κάνει αρκετές εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας, έξι και αυτή θα είναι η έβδομη και όγδοη έκθεση που κάνουμε για το θέμα αυτό. Ήταν εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας, αλλά μας αγνοούν παντελώς. Δεν βοηθά καθόλου αυτό που κάνουμε. Στις προηγούμενες εκθέσεις προσπαθούσαμε να προτείνουμε ε, να δημιουργηθούν οι κατάλληλε προποθέσει για διοργανική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρχει πλήρης δημοκρατική συμμετοχή. Μπορεί να χρειάζεται και αλλαγή της συνθήκης. Αλλά χωρίς αλλαγή της συνθήκης και πάλι μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Και εγώ πραγματικά εξακολουθώ να μην μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μας υποστηρίζει το ΕΛΚ. Γιατί δεν υποστηρίζεται τη δημοκρατική συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να μου απαντήσει και να το συζητήσουμε αυτό πριν ψηφίσουμε. Να σας πω επίσης ότι υποστηρίζω ε, πλήρως τις παρατηρήσεις για να έχουμε το scoreboard, αυτό τον ε, κατάλογο των αποτελεσμάτων ε, και την κοινωνική διάσταση. Δυστυχώς αυτό δεν υποστηρίστηκε ε, ούτε καν από τους σοσιαλιστές και πραγματικά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μια διατύπωση την οποία θα μπορούσαν να δεχτούν οι περισσότεροι γιατί θεωρώ ότι είναι ζωτική σημασία όταν υπάρχει ένας κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων να ε, αποφέρει αποτελέσματα. Να μην είναι απλώς στατιστικά στοιχεία τα οποία μας δείχνουν πόσο φρικτά είναι τα πράγματα. Τι ξέρουμε. Ε, θέλουμε απλώς να γίνει κάτι γι' αυτό. Και μια τελευταία παρατήρηση θα πρέπει αφενός να καλωσορίσουμε το γεγονός ότι ε, γίνεται έρευνα για τα πλεονάσματα της Γερμανίας, αλλά θα πρέπει να επικρίνουμε και την παρατήρηση του Μπαρόσο ο οποίος είπε αμέσως ότι ναι μεν, αλλά αν το πλεόνασμα είναι επιζήμιο, δεν θα υπάρξει πρόστιμο για τη Γερμανία. Κάτι το οποίο υποσκάπτει την ίση μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών και υποσκάπτει και την ίδια τη διαδικασία της ισορροπίας. Διότι το σκεπτικό ήταν ότι θα υπάρχει ισορροπία, εξισορρόπηση της ευρωπαϊκής οικονομίας προς όφελος όλων και τα πλεονέσματα μπορεί να είναι εις βάρος αυτής της ισορροπίας εξίσου με τα ελλείμματα. Ελπίζω λοιπόν να υποστηρίξουν και οι υπόλοιποι μια τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Χάρκιν. Ε, είχαμε εδώ μια μικρή συζήτηση σχετικά με το γερμανικό πλεόνασμα. Δεν συμφωνούμε απολύτως μεταξύ μα, βέβαια. Ευχαριστώ τον κύριο Κουτιέρες Πριέτο για την έκθεσή του. Δεν ε, θα μπω σε πολλές ε, λεπτομέρειες, ε, διότι τώρα αρχίζω να ασχολούμαι με το θέμα, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ καλές ιδέες εδώ. Ιδιαίτερα την αρχή του front-loading να ε, ξεκινήσει το Ταμείο από το 2014 και μετά. Ε, αυτό νομίζω μπορεί να βοηθήσει κάποιες οικονομίες. Ε, μια παρατήρηση για τις δουλειές ποιότητας, τις θέσεις εργασίας ποιότητας. Κάποιοι θέλουν να εργαστούν με μερικό ωράριο. Δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τον όρο αυτόν. Ξέρω ότι υπάρχουν διάφοροι, ε, διάφορα είδη μερικής απασχόλησης ε, και πρέπει να είναι σαφές το τι συζητάμε εδώ πέρα. Νομίζω ότι αν είναι καθαροί οι όροι ε, θα δούμε ότι συμφωνούμε μεταξύ μας. Επίσης όσον αφορά τις προγνώσεις για ανάπτυξη είναι κάτι που έχω αναφέρει στο παρελθόν καθώς και πολλοί άλλοι. Θα πρέπει να βρούμε πιο ακριβώς ακριβή τρόπο ε, πρόγνωσης. Ε, άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπε η κυρία Λόπε Φοντάνια, μίλησε για την Ισπανία και για ε, την δημοσιονομική εξυγίανση. Δεν μπορώ να μιλήσω για την Ισπανία, διότι δεν γνωρίζω αρκετά για το θέμα. Αλλά αν δει κανεί τι λέει το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και άλλοι, οι θέσει του είναι κάπως, έχουν πιο πολλές αποχρώσεις. Υπάρχει ο κίνδυνος ε, αποπληθωρισμού και ε, αυξανόμενων ανισορπιών ε, εντός της Ευρώπης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να μπορεί να πει ότι αυτό δεν συμβαίνει. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο η δημοσιονομική εξυγίανση, ότι αυτό είναι κάτι καλό και ότι όλα τα άλλα πράγματα είναι κακά. Ξέρω ότι και στη δικά σας έκθεση μιλήσατε για ευελιξία. Το χρειαζόμαστε αυτό. Νομίζω ότι μπορεί να χρειαστούμε και κάποια στοιχεία ακόμα. Τέλος, ε, η πρόεδρος ε, μας ε, προειδοποίησε και νομίζω ότι είναι πολύ καλές οι συμβουλές της διότι έχουμε τη διαδικασία της συναπόφασης και θα πρέπει να μπορούμε να επηρεάσουμε τη διαδικασία περισσότερο από το απλά να νιώθουμε καλά για το τι έχουμε κάνει. Αλλά ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα και όσον αφορά τη δημοκρατική νομιμότητα απέχουμε ένα εξάμεινο από ευρωεκλογέ. Εάν οι άνθρωποι που θα πρέπει να μας ψηφίσουν νιώθουν ότι δεν έχουμε λέγει στα όσα γίνονται, ε, τότε δεν, μάλλον δεν θα πρέπει να ζητάμε την ψήφο τους. Thank you so much. I would like... Η Edith Bauer. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ε, κάνω μία σύντομη παρατήρηση. Πριν περίπου 20 λεπτά η Eurostat εξέδωσε, κοινοποίησε νέες στατιστικές ε, για την φτώχεια. Ο τίτλος είναι το 2012 το 1 τέταρτο του πληθυσμού βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή ε, κοινωνικού εξοπλισμού, κάτι που ε, αντιστοιχεί σε 125 εκατομμύρια ανθρώπων. Ε, είναι τεράστιο νούμερο αυτό, δεδομένου ότι μιλούσαμε για 80 εκατομμύρια όταν υιοθετήθηκε η στρατηγική 2020. Έχω λοιπόν την εντύπωση πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε πιο σοβαρά το θέμα αυτό από ό,τι μέχρι τώρα. Θα ήθελα επίσης να συμφωνήσω με την θέση του εισηγητή σχετικά με τα χρέη του πληθυσμού, διότι νομίζω ότι είναι ε, ένα θέμα ε, το οποίο υποτιμάται μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ. Υπάρχει ένας άλλος που θέλει το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Καλώς, οπότε ο εισηγητής. Καταρχάς, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και για τα στοιχεία που συνέβαλαν. Μέσω των ομιλιών τους, τους στην συμπερίληψη. Προσπαθούμε λοιπόν να συμβάλλουμε στη συζήτηση και να προωθήσουμε κάποιες αλλαγές. Συμφωνώ με την κυρία Λόπε Φοντανέ ότι η διαδικασία δημοσιονομικής εξυγένσης αλλάζει την μακροοικονομική κατάσταση. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν θετικά τμήματα, αλλά τα θετικά αυτά έγιναν λόγω της δικής μας παρέμβασης, διότι ε, ε, καταφέραμε να επιβάλλουμε κάποια ελαστικοποίηση αυτής της διαδικασίας. Βεβαίως πρέπει να μειώσουμε τα ελλείμματα, αλλά αυτό που πάντα προσπαθούμε να τονίσουμε στη συζήτηση είναι με ποια ταχύτητα και επίσης την άλλη πλευρά, την άλλη όψη του νομίσματος. Δηλαδή πρέπει να τονώσουμε την ανάπτυξη και κυρίως τη δημιουργία απασχόλησης. Αυτό που λέμε στην έκθεση. Τι λέμε. Όπως αναγνώρισε και η Κομισιόν στις ετήσιες προβλέψεις είναι ότι πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση ε, της, ε, του ρυθμού εξυγένσης. Άρα θεωρούμε ότι όταν ξεκίνησε η διαδικασία υπήρχε ήδη κάποια λάθος αντίληψη που δεν θα πρέπει να συνεχιστεί. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που λένε εάν ήταν πιο διαφοροποιημένη η διαδικασία δημοσιονομικής εξυγίανσης θα μπορούσε να έχει μειωθεί η απασχόληση κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο. Και ξέρετε τι σημασία έχει η απασχόληση για να αντιμετωπιστεί μια τόσο σκληρή κρίση. Θεωρώ λοιπόν, συμφωνώντας με την κυρία Κορνέλισεν και την κυρία Άρκιν, ότι είναι αναγκαίο να συνεχίσουμε να τονίζουμε το δημοκρατικό τμήμα αυτής της έκθεσης, γιατί μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή και τα εθνικά κοινοβούλια και οι κοινωνικοί εταίροι. Διότι οι πολιτικές που υιοθετούνται στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής δεν συμπεριλαμβάνει επαρκώς τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων, των πολιτών. Ιδιαίτερα ελπιρό είναι ότι πολλά κράτη-μέλη δεν είχαν συζητήσει τα εθνικά τους ε, προγράμματα σύγκλησης και σταθερότητας ούτε με τους κοινωνικούς εταίρους, ούτε στα πλαίσια των Εθνικών Κοινοβουλίων όταν αποφάσισαν το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Στόχος μας λοιπόν είναι να διορθώσουμε αυτή την έλλειψη. Για το εμπορικό πλεόνασμα, συμφωνώ με την κυρία Κορνέλσεν. πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τον πιο κατάλληλο τρόπο, πρέπει να τονώσουμε την εσωτερική ζήτηση, την απασχόληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τίθεται και το θέμα της ποιότητας της απασχόλησης. Δεν έχω αντίρρηση εγώ σε συμβόλαια συμβάσεις περιορισμένου χρόνου. Αλλά σε πολλά μέρη της Ευρώπης, ξέρετε, αυτά τα συμβόλαια δεν ε, υπογράφονται εθελουσίως από τις δύο πλευρές. Οι εργαζόμενοι τα υπογράφουν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Έχουν γίνει και μελέτες από κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς που τονίζουν ότι αυτά τα συμβόλαια μερικής απασχόλησης καλύτερα στην ουσία οδηγούν τους εργαζόμενους να δουλεύουν όλη τη μέρα και να πληρώνονται σαν να δουλεύουν μόνο μερικώς. Αυτό πρέπει να το αναλύσουμε. Βεβαίως, σε ορισμένες περιοχές είναι πολύ λιγότερα τα συμβόλαια μερικής απασχόλησης από ότι είναι ο μέσος όρος στην Ευρώπη. Αυτήν την ε, ανισορροπία πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Κατά τα υπόλοιπα, ευχαριστώ όλους τους ομιλητές Έχουμε λίγο χρόνο, όπως είπε και η κυρία Φοντανέ, αλλά μπορούμε να κάνουμε καλή δουλειά. Χρειάζεται λοιπόν πολλή ε, διάλογος, αν και πρέπει να εργαστούμε ταχύτατα, αλλά πρέπει, όπως είπε και η κυρία Κορνέλσεν, αυτή πρέπει να είναι η τελευταία έκθεση, η προηγούμενη δηλαδή, Πρέπει να είναι η τελευταία έκθεση η οποία δεν εισακούστηκε. Πρέπει λοιπόν να επιτύχουμε περισσότερη συνένεση για να εισακουστούν οι προτάσεις μας Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, σας ευχαριστώ. Παρά τις διεκδικήσεις σας δεν θα αλλάξουμε την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. 10 Δεκεμβρίου στις 12 η ώρα εκπνέει η προθεσμία. Θα τις εξετάσουμε στις 17 Δεκεμβρίου, 22 Ιανουαρίου θα τα συζητήσουμε, θα συζητήσουμε τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε την επομένη 23 Ιανουαρίου και εκείνη την ίδια εβδομάδα 20, 21 και 22 Ιανουαρίου θα έχουμε τις ημέρες διαβουλεύσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια για το θέμα αυτό. Ε, ολοκληρώσαμε λοιπόν με το σημείο αυτό στην σε διάταξη. Συνεχίζουμε. Στο σημείο 4 όπου θα πρέπει να εξετάσουμε τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου που έγινε στις 27 Νοεμβρίου για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για τη διοργάνωση δειγματοληπτικής έρευνας σχετικά με το οργανωτικό δυναμικό της κοινότητας. Να δώσω το λόγο στην Τατιάνα Ζανόκα, την ησυχήτριά μας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, διότι υπήρξε μία παρανόηση για την ώρα που θα εξεταστεί η έκθεση. Έπρεπε να βρίσκομαι σε τρία σημεία ταυτόχρονα. Ήμουν στους συντονιστές στην Επιτροπή Αναφορών σήμερα το πρωί. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν. Όσον αφορά τώρα την έκθεση ή μάλλον τον τριμερή διάλογο. Καταρχάς να ευχαριστήσω την Πρόεδρο για τη διεξαγωγή του τρομερού διαλόγου και ελπίζω να συνεισφέρει πολύ στη συμφωνία. Ευχαριστώ βεβαίως και το προσωπικό της Επιτροπής Απασχόλησης για τη βοήθειά τους. Θα σταθώ σε ένα βασικό σημείο της συμφωνίας πλέον μεταξύ του Συμβουλίου και του κειμένου της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της θέσης του Κοινοβουλίου. Αυτό αφορά ε, τα ad hoc ερωτηματολόγια για αυτή τη δειγματολογική έρευνα. Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να γίνονται αυτά μέσω πράξεων κατεξουσιοδότηση. Ναι, το Κοινοβούλιο ενέκρινε αυτή την αρχική πρόταση και δεν κατέθεσε τροπολογίες στο τμήμα αυτό για την τροποποίηση του κανονισμού για την έρευνα για το εργατικό δυναμικό, αλλά το Συμβούλιο πρότεινε να έχουμε εκτελεστικές πράξεις. Και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να καθορίσει τους δείκτες ε, ε, για το, η έρευνα και έτσι θεωρούν ότι τα κράτη-μέλη δεν θα έχουν λόγο, θα επιβάλλονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των ε, πράξεων κατεξουσιοδότηση για όλες τις μεταβλωτές αυτής της έρευνας. η θέση μας σε όλη τη διάρκεια αυτού του διαλόγου ήταν ότι επιμένουμε να έχουμε πράξη καταξουσιοδότηση που δίνει τη δυνατότητα και στο Κοινοβούλιο να παρέμβει όταν λαμβάνει προτάσεις για αυτά για αυτές τις ad έρευνες ε, και αυτά τα συγκεκριμένα μοντέλα, κυρίως διότι αυτά τα μοντέλα έχουν πολιτικό περιεχόμενο. Τα τελευταία ε, ήταν για την ανεργία των νέων. Το 2014 θα έχουμε κάποια ε, ερωτηματολόγια για την ε, απασχόληση των μεταναστών, ε, τα επαγγελματικά προσόντα και ούτω καθεξής. Από τις τελευταίες πληροφορίες που έχω από το Συμβούλιο, θα κάνουν μια συμβαστική πρόταση. Θέλουν να υπάρχει μια επιτροπή του Συμβουλίου που θα εξετάζει τις προτάσεις αυτές για αυτά τα ad hoc ερωτηματολόγια, να υπάρχουν δηλαδή εκπρόσωποι των κρατών μελών και να έχουν αυτοί το δικαίωμα να καθορίσουν τον κατάλογο των μεταβλητών. Και όλες οι υπόλοιπες παράμετροι να περνούν με πράξη κατεξουσιοδότηση όπως ε, προτείνεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα ad hoc ερωτηματολόγια. Αυτά λοιπόν ενημερωτικά. Για όσους συμμετέχουν στον τριμερή διάλογο, στις 17 Δεκεμβρίου θα γίνει ο δεύτερος τριμερός διάλογος. Δεν έχουμε ακόμα κάποια γραπτή πρόταση από πλευρά Συμβουλίου για τη συμβιβαστική τους πρόταση. Θα πρέπει να την εξετάσουμε πρώτα και να προετοιμαστούμε φυσικά για τον τριμερή διάλογο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πλήρης ε, αναφορά για τα όσα κάναμε και δείχνει πόσο καλές είναι αυτές οι διοργανικές μας σχέσεις. Υποχρεωθήκαμε να στείλουμε επιστολή στο Συμβούλιο για να διευκρινίσουμε το επίπεδο φιλοδοξίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλει κάποιος το λόγο? Δεν βλέπω κάποιον. Καλό κουράγιο λοιπόν και σε εσά και σε εμά για τον επόμενο τριμερή διάλογο, ο οποίο, όπως μας είπατε κι εσείς θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου. Ολοκληρώσαμε λοιπόν με αυτό το σημείο της σας διάταξης και περνάμε τώρα στο σημείο 12. Εδώ έχουμε την νομοθετική πρόταση για την ενισχυμένη συνεργασία των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης. Έκθεση του κυρίου Φεντερικ Νταρντά στον οποίο δίνω αμέσως το λόγο για την εξέταση των συμβιβαστικών τροπολογιών και ζητώ συγγνώμη γιατί θα πρέπει να ε, αποχωρήσω και θα δώσω το λόγο ε, την Προεδρία στην κυρία Edith Bauer, η οποία είναι η γυρεότερη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας αφήνω να κάνετε την αλλαγή. Quelques mots sur ces compromis. Δύο λόγια λοιπόν για αυτές τις συμβαστικές προτάσεις για την ενισχυμένη συνεργασία των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης. Δεν θα υψέλθω στην ουσία της πρότασης, διότι το είχαμε συζητήσει αρκετές φορές εδώ στην Επιτροπή μας. Θα σας πω δύο λόγια μόνο για τις συμβαστικές τροπολογίες. Κατατέθησαν 17 συμβαστικές τροπολογίες και ίσως θα υπάρξει και μια 18η. για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις περισσότερες από τις τροπολογίες οι οποίες υπευλήθησαν. Ε, ε, Είμαστε σε κάποιες επαφές για να τελειοποιήσουμε λίγο τη διατύπωση σε αυτές τις τροπολογίες. Δεν θα, θα αναφερθώ ε, σε όλες, ε, θα αναφερθώ σε τέσσερα θέματα. Το πρώτο θέμα αφορά τις τροπολογίες ε και ν και η εκπροσώπηση ε, σε εθνικό επίπεδο των ε, μελών αυτών. Ε, θέλουμε να έχουμε αναπληρωτές εδώ και θέλουμε να διατηρήσουμε και μία ψήφο αναχώρα στο Συμβούλιο αυτού του δικτύου. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο προκύπτει από κάτι το οποίο έχει γίνει σε ένα άλλο ζήτημα ε, για την πρωτοβουλία για τους νέους. Δεύτερον, συμβαστική τροπολογία M, συνεργασία του δικτύου με άλλους αρμοδίους σε θέματα πολιτικής απασχόλησης. Και εδώ θεωρούμε ότι είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία, διότι είναι χρήσιμη και ε, υπάρχουν αρκετοί εταίροι, γι' αυτό ακριβώς αναφέρονται και αυτοί στη συμβαστική πρόταση. Επιμένουμε λοιπόν στο γεγονό ότι αυτή η συνεργασία θα πρέπει να γίνεται με πρωτοβουλία του ίδιου του δικτύου, ανάλογα με τα θέματα τα οποία τους απασχολούν. Τρίτον, συμβαστική τροπολογία όμικρον για τις πράξεις κατεξουσιοδότηση. Εδώ Έγινε μια συζήτηση μεταξύ μας για να δούμε μέχρι ποιου σημείου μπορούμε να, δούμε, να έχουμε χώριση εξουσιών και μάλιστα σε ποιον. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και το σημαντικό είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα χάσει τελείως την επιρροή του ως προς τη διαδικασία. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε μια συμβαστική πρόταση βάσει τις οποίες κάποιες από τις αποστολές του δικτύου θα είναι με πράξεις εκτελεστικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, θα είναι αρμοδιότητα του δικτύου. Θεωρώ ότι το Συμβούλιο και θα έχουμε και την ευκαιρία ε, να το συζητήσουμε το θέμα αυτό στον τριμερή διάλογο ε, προτιμά περισσότερο εκτελεστικής πράξης αλλά θα πρέπει και εμείς να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε κάποιο ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέταρτον, Κάτι το οποίο δεν περιλαμβάνεται ακόμα στο έγγραφο το οποίο συζητούμε για τις συμβαστικές προτάσεις. Το κατά πόσον θα είναι υποχρεωτική ή εθελοντική η συμμετοχή στο δίκτυο των ε, δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης των διαφόρων κρατών μελών. Κατ' εμέ, διαβάζοντα την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν προφανέ ότι ήταν υποχρεωτική η συμμετοχή και από εκεί και πέρα θα μπορούσε να υπάρχει θελοντική ε, συμμετοχή κάποιων άλλων, αλλά από ό,τι φαίνεται η θέση του Συμβουλίου είναι διαφορετική. Γι' αυτό ακριβώς και εγώ προτείνω να υπάρξει μια συμβιβαστική τροπολογία που θα μπορούσε να βασίζεται στην τροπολογία 44 και να πούμε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, τις οποίες ανα, καθορίζει κάθε χώρα. Δηλαδή κάθε χώρα θα συμμετέχει υποχρεωτικά ε, σε αυτό το συμβούλιο, σε αυτό το δίκτυο. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα τα οποία ήθελα να θέσω εδώ για να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Δύο ζήτησαν το λόγο, ο κύριος Πέκερ και ο κύριος Πένιον. Κύριε Πέκερ, είναι τιμή μου να μπορώ να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι προνόμιο για μένα να μιλώ υπό την Προεδρία σας. Θα ήθελα και εγώ να πάρω το λόγο, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ε, θα ήθελα να τονίσω την ε, εκτίμησή μου για τη συνεργασία με τον ε, εισηγητή που ήταν ε, πάρα πολύ επαγγελματική, πάντα εντός θέματος. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει ότι υπάρχουν δύο θέματα για τα οποία δεν είμαι ικανοποιημένος και θέλω να αναφερθώ στην συμβαστική τροπολογία N, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον θεσμικό τομέα Κάθε κράτος μέλος ε, έχει σχεδόν πάντα εκπρόσωπο σε οποιοδήποτε φόρουμ. Με την διατύπωση αυτή, ε, το θέμα αυτό παίρνει διαστάσεις τις οποίες δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Σκέφτομαι τις χώρες που έχουν διάφορες περιφερειακές ε, ε, ε, διοικήσεις για την αγορά εργασίας και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν βελτιώνει την ποιότητα των εργασιών στα συμβούλια αυτά. Θα πρέπει να το σκεφτούμε λοιπόν να έχουμε Το να έχουμε έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και έναν αναπληρωτή, ε, αυτό ε, νομίζω ότι είναι απολύτως επαρκές. Ε, αν έχουμε περισσότερους, αυτό θα είναι εις βάρος της δουλειάς. Επίσης, οι επιθεωρήσεις εργασίας έχουν να παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτική απασχόληση, όχι όμως στην πολιτική της αγοράς εργασίας, αλλά στην καταπολέμηση της ανεργίας. Στον τομέα αυτών λοιπόν ε, δεν έχουν ε, αρμοδιότητες ούτε γνώσεις. Δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν οι επιθεωρήσεις εργασίας. Τρίτον, ο κύριος Δαρντέν το ανέφερε αυτό. Είναι το θέμα της υποχρεωτικής ε, ή προαιρετικής συμμετοχής. Συμφωνώ απολύτως με την πρόταση του εισηγητή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπένιον, έχετε το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, δουλειά του πάνω στο θέμα αυτό. Δεν ήταν πάρα πολύ επίμαχο το θέμα αυτό. Νομίζω θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβασμούς στα περισσότερα θέματα. Έχουμε κάποιες δυσκολίες με τη συμβαστική τροπολογία M μέχρι στιγμής. Μη θα προτιμούσα να, λέμε regular αντί για occasional, ε, τακτικό αντί για ε, συχνό, αλλά το, το, και ο τακτικός ε, δεν χρειάζεται να είναι συχνός. Αλλά ε, δεν είναι και ad hoc. Επίσης, ανησυχούμε λίγο σχετικά με τους εκπροσώπους. Οι κοινωνικοί εταίροι δεν είναι πάντα οι κατάλληλοι φορείς ιδιαίτερα όχι όταν ε, μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις. Ε, συχνά οι μικρές επιχειρήσεις όσον αφορά τους εργοδότες και τους εργαζομένους ε, είναι τελείως διαχωρισμένες από τους κοινωνικούς εταίρους. Αυτά όμως είναι περισσότερο επιμέρους. Το σημαντικό θέμα είναι στη συμβαστική τροπολογία I. θεωρώ ότι είναι σωστό να χρησιμοποιούμε τον όρο κοινωνικό dumping σε νομοθετικό κείμενο, διότι δεν έχουμε ορισμό ουσιαστικά επιβάλλουμε στο δίκτυο έτσι μια υποχρέωση με την οποία δεν μπορεί να συμμορφωθεί. Παρότι λοιπόν δεν έχουμε πρόβλημα με τη χρήση του όρου κοινωνικό ντάμπινγκ σε άλλα κείμενα, ε, δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε ένα νομοθετικό κείμενο. Τη στιγμή που δεν υπάρχει σαφής και γενικά αποδεκτός ορισμός. Επίσης, όσον αφορά τον ορισμό, ε, το, τη συμβαστική τροπολογία Q, ε, δεν νομίζουμε ότι είναι απαραίτητο, γιατί απλά επαναλαμβάνουμε το άρθρο 3.1α. Ε, πάντως νομίζω ότι έχουμε χρόνο να ε, καταλήξουμε σε συμβασμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν θέλει το λόγο. Κύριε Νταρντά, θέλετε να συνοψίσετε. Avec Βεβαίως. Οπότε, για την παρέμβαση του κυρίου Μπέκερ και τη συμβαστική πρόταση ένανι. Τον κίνδυνο δηλαδή να υπάρξουν πολλοί αναπληρωματικοί και να είναι δύσκολη λειτουργία του οργάνου αυτού. Καταλαβαίνω την πρότασή του και σε έναν βαθμό να συμφωνήσω μαζί του, να βρούμε μια τύπωση πιστεύω, θα τα καταφέρουμε. Ίσως θα μπορούσαμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αναπληρωτών. Ε, ίσως να αρκεί ένας, μ, ίσως να είναι λίγοι μόνο ένας αναπληρωτής. Το βασικό είναι ο ή οι λίγοι αναπληρωτές να μπορούν να συμμετέχουν στις συζητήσεις και να μην αντικαθιστούν απλώς όταν λείπει το τακτικό μέλος, να μπορούν να παρακολουθούν τη συζήτηση όλη τη διαδικασία. Θεωρώ ότι αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, για την επιθεώρηση εργασίας. Το άλλο θέμα που αναφέρατε. Ναι, το σκέφτηκα και συμφωνώ μαζί σας. Η επιθεώρηση εργασίας δεν θα πρέπει να συμμετέχει στο δίκτυο ως οργανισμός. Μπορούν να συμβάλλουν σε κάποιες φάσεις, σε μια γενικότερη εξέταση κάποιων θεμάτων που θα ξεκινήσουν οι δημόσιοι οργανισμοί απασχόλησης θα μπορούσαν για παράδειγμα να δώσουν τη γνώμη τους ε, σε κάποια συζήτηση κάποιου συγκεκριμένου θέματος αλλά δεν χρειάζεται να ανήκουν στο δίκτυο. Θα βρούμε πιστεύω και για το ζήτημα αυτό ένα συμβασμό. Σας ευχαριστώ ε, επίσης που στηρίζεται τον υποχρεωτικό χαρακτήρα που νομίζω ότι είναι σημαντικός. Για τις παρατηρήσεις του κυρίου Μπένιον. Για τη συμβαστική πρόταση M, Συμφωνώ. Το περιστασιακό δεν είναι ο καλύτερος όρος. Δεν είναι καλό να βάλουμε περιστασιακό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό είναι να γίνεται με πρωτοβουλία του δικτύου. Να βάλουμε τακτικά ή να μην βάλουμε κανέναν όρο. Ούτε τακτικά, ούτε περιστασιακά. Και να πούμε απλώς κάθε φορά που χρειάζεται με πρωτοβουλία και νομίζω πως τακτικά θα είναι αναγκαίο για να μην υπάρχει φορμαλισμός σε αυτό το επίπεδο. Αυτά για την συμβαστική πρόταση μη. Για το ποιοι εκπροσωπούν τους εργαζόμενους, να βάλουμε κοινωνική εταίρη δεν είναι δική μου η πρόταση. Θα μπορούσα να την αποδεκτώ, αλλά ίσως πρέπει να το ξανασυζητήσουμε για να μην αποκλείσουμε κάποιες καταστάσεις. Το βασικό είναι να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Αντίθετα, για την συμβαστική τροπολογία I, Ι, είναι σημαντικό εφόσον θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ανεργία και στόχος των ε, υπηρεσιών απασχόλησης είναι η καταπολέμηση της εργασίας. Εφόσον λοιπόν μιλάμε για αυτό το θέμα, πρέπει να αναφερθούμε στο κοινωνικό ντάμπινγκ, μπορεί να μην υπάρχει επίσημος ορισμός, αλλά ε, το θέμα αυτό προκαλεί ανεργία σε κάποιες περιοχές. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε το θέμα του κοινωνικού ντάμπινγκ. Το θεωρώ όχι μόνο χρήσιμο αλλά και αναγκαίο. Πιστεύω λοιπόν ότι τουλάχιστον η έννοια πρέπει να διατηρηθεί. Μπορούμε να το συζητήσουμε για τη διατύπωση. Ευχαριστώ νομίζω ότι έτσι απάντησα αυτά τα θέματα που έθεσαν οι συνάδελφοι. Αλλά έχουμε και κάποιες μέρες ακόμη για να ε, επεξεργαστούμε περαιτέρω το κείμενο μέχρι τη Δευτέρα νομίζω. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα είναι τη Δευτέρα, όπως είπε και ο κύριος Νταρντέν. Στην Ολομέλεια υποθέτω ότι θα είναι στην ημερήσια διάταξη του Μαρτίου ή του Απριλίου. Και τώρα να περάσουμε στο 13. Πάλι ο κύριος Πριέτο. Η μέρα σας σήμερα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ που είναι η μέρα μου. Δύο σχόλια μόνον. Ένα να ευχαριστήσω τους υπόλοιπες συναδέλφους, τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες, διότι πάντα είναι διατεθειμένοι να καταλήξουν σε συμφωνία. Έχουμε συζητήσει ήδη τις τροπολογίες την προηγούμενη εβδομάδα και είδαμε ότι υπήρχε ευρύτατη συνένεση για την έκθεση με κάποιες μικρές διευκρινήσεις, τις οποίες νομίζω ότι έχουμε συμπεριλάβει σε γενικές γραμμές τις τρεις συμβαστικές προτάσεις που καταθέσαμε. Θα ήθελα απλώς ε, να τονίσω ότι είναι σημαντικό το γεγονό ότι έχουμε αυτή την έκθεση, διότι οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις μπορούν να προσδώσουν μεγαλύτερη σταθερότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία και νομίζω ότι αυτό μας οδηγεί στη σωστή κατεύθυνση για να διορθώσουμε σφάλματα των περασμένων δεκαετιών και επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο ε, συνεισφέρουμε εμείς ως Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, να ευχαριστήσω τους και συζητητές και για τις τροπολογίες τους και για τη συνεισφορά, επίσης και για τις συμβιβαστικές προτάσεις τις οποίες καταλήξαμε και τη διάθεσή τους να καταλήξουμε σε συμφωνία και θεωρώ ότι θα μπορέσει ε, τελικώς να προκύψει μια καλή έκθεση η οποία θα μπορέσει να βοηθήσει αυτή τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση η οποία θα βελτιώσει την ε, Ευρωζώνη. Τίποτα άλλο, να πω και πάλι ότι ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν, ε, κυρίως ε, τους και ηγετές για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πριέτο. Ο κύριος Ογκούριαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Είναι καλή έκθεση. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Καλή δουλειά. Και θα υποστηρίξουμε τις συμβαστικές ε, τροπολογίες. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλα προβλήματα με την έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Όχι. Να σας υπενθυμίσω ότι θα ψηφίσουμε τη Δευτέρα στην έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Απασχόλησης στο Στρασβούργο και στην Επιτροπή ΕΚΟΝ η ψηφοφορία θα γίνει στις 20 Ιανουαρίου και κατά πάσα πιθανότητα θα συμπεριληφθεί στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου το θέμα αυτό. Και τώρα θα περάσουμε στο σημείο 14 της ημερησίας διάταξης και να σας ενημερώσω εγώ λίγο για το πώς έχει κατάσταση για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων την κατάσταση αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ορισμένες φορές μας δίνεται η αίσθηση ότι ακόμα και σε σύγκριση με τον κανονισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θέλουν να περιορίσουν το πεδίο εφαρμογής αλλά ελπίζω ότι θα έχουμε το να, να διατηρήσουμε τις θέσεις μας. Δεν θα είναι εύκολο. Όλοι όσοι συμμετέχουν γνωρίζουν ότι πραγματικά δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ακόμα δεν έχουμε ε, κάποια απάντηση από πλευρά Συμβουλίου ως προς τις προτάσεις μας. Παραδείγματος χάρη για την ε, δυνατότητα διαμονής, ε, το να συμμετέχουν ή να αναφέρονται οι κοινωνικοί εταίροι συνολικά, όπως επίσης και κάποια άλλα θέματα. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η διαπραγμάτευση. Ελπίζω να γίνει ένας έκτακτος τριμερής διάλογος την επόμενη εβδομάδα και ελπίζουμε επίσης ότι στις 18 ή στις 16 Δεκεμβρίου θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Όλα αυτά βέβαια είναι ελπίδες, διότι οι διαπραγματεύσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες και προχωρούν πάρα πολύ αργά. Θέλει κάποιος το λόγο, ο κύριος Θέρκας. Ναι, ευχαριστώ κύριε Μπάουερ. Να υπενθυμίσω απλώς τους συναδέλφους, ή μάλλον καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη γιατί ο κύριος Κρίστενσεν είναι σε μια επίσημη συνεδρίαση με ε, την κυβέρνησή του και δεν μπορεί να είναι εδώ και για να μιλήσω για τα δύο θεμελιώδη ζητήματα τα οποία γνωρίζετε εσείς κυρία Μπάουερ διότι ε, τον ίδιο αγώνα δίνουμε αλλά να τονίσω ότι για τους σοσιαλιστές είναι άκρος απαραίτητο και πρέπει να το πείτε στο Συμβούλιο ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε τίποτα κυρίως το άρθρο 4 το οποίο να απειλεί τις ε, εθνικές παραδόσεις για τις συλλογικέ συμβάσεις και την νομιμοποίηση και την ενεργητική και την παθητική όσων ε, προσυπογράφουν τις συλλογικέ συμβάσεις. Η Ευρώπη πρέπει να συμμορφούνται προς τις συνθήκες και στις συνθήκες υπάρχει υποχρεωτικό σεβασμός στην αυτονομία των ε, κοινωνικών εταίρων και τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι εργασιακές σχέσεις σε εθνικό επίπεδο δεν είναι δυνατόν να αλλάξει με μάλιστα περίεργο τρόπο η νομοθεσία των κρατών μελών στα θέματα αυτά. Ε, είτε έχουμε δημοψήφισμα, είτε υποχρεωθές είτε οτιδήποτε, θα πρέπει να γίνεται σεβαστό ότι υπάρχει σε κάθε χρόνο και είναι ιστορικό και υπάρχει στην ε, οργάνωση των εργασιακών σχέσεων. Αυτό είναι το βασικό, το άρθρο 4 και επίσης να τονίσω και ότι σε κάποια αιτιολογική σκέψη υπάρχει ένα στοιχείο που δημιουργεί σύγχυση σε σχέση με το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να καλύπτονται, να έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Ναι, είναι διαφορετικό, αλλά όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να καλύπτονται σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορεί να υπάρχει κάποια μαύρη τρύπη από την οποία θα χαθούν συγκεκριμένε ομάδες εργαζομένων μέσω ε, μιας διατύπωσης η οποία θα είναι τόσο συγκεχημένη που θα δώσει τη δυνατότητα να υπάρχουν μια σειρά από παρερμηνίες και να καταλήξουν όλες αυτές οι υποθέσεις στο δικαστήριο θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι συλλογικέ συμφάσεις και το πεδίο εφαρμογή ε, της οδηγίας αυτής ε, και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλίνει από αυτό το κανονισμό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μπένιον. Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις επί της Γενικής Αρχής. Ε, δεν συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις αυτές, οπότε είναι δύσκολο να γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να θέσουμε ένα όριο όσον αφορά την ελεύθερη κινητικότητα των εργαζομένων, ιδιαίτερα όταν αυτή γίνεται για λόγους εργασίας. Αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις ε, στην ε, απόσπαση Μπορεί να επανέλθουμε σε αυτό την ε, επόμενη εβδομάδα, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν τομείς όπου υπάρχουν ανησυχίες και τομείς όπου δεν είναι σαφές στα κράτη-μέλη ε, τι γίνεται με την ελεύθερη κινητικότητα και με την μεταφορά δικαιωμάτων. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ. Μια σύντομη παρατήρηση. Σχετικά με τις δύο αυτές παρεμβάσεις. Όσον αφορά το άρθρο 4, προσπαθούμε να διατηρήσουμε τη θέση μας. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Κάτι που μάθαμε από τις διαπραγματεύσεις αυτές είναι ότι σε τέτοιε περιπτώσεις όπου οι διαφορέ οφείλονται σε διαφορετικές ε, νομικές παραδόσει. είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρουσιάσετε και στο Συμβούλιο αυτή η διαφορά. Ε, εάν οι εκπρόσωποι των ε, χωρών αυτών συμφωνήσουν με το κείμενο, είναι πολύ δύσκολο να υπερασπιστούμε μια τέτοια θέση, διότι το ερώτημα που έθεσε η Προεδρία ήταν γιατί δεν ακούστηκε αυτό στο Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί κανείς παρά να συμφωνήσει. Ε, αυτό θα πρέπει να ενδιαφέρει όχι μόνο εμάς, αλλά και τη συγκεκριμένη χώρα. Όσον αφορά την παρατήρηση του συναδέλφου Μπένιον, θα ήθελα να πω ότι η οδηγία αυτή κατά κάποιο τρόπο είναι απλά μια οδηγία εφαρμογής ήδη ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα αυτών. Δεν αφορά την απόσπαση εργαζομένων, αυτοί αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής. ούτε θεσπίζονται εδώ νέα δικαιώματα. Ακόμα και το πεδίο εφαρμογή ε, είναι το ίδιο. Γι' αυτό νομίζω ότι ε, απλά συμβάλλει στο να γίνει πιο καθαρή η κατάσταση τώρα από την αυτή, ε, στο μέλλον από την αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε την ε, ημερήσια διάταξη. Η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα στις 7.30 στο Στρασβούργο και μετά στις 17 Δεκεμβρίου το απόγευμα. Κάτι ασυνήθιστο. Έχουμε συνεδρίαση μόνο το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενεργό συμμετοχή σας. Ε, καλό Σαββατοκυριακό.